Κυρία Πάκ, για τη δική σα έκθεση έχετε να πείτε κάτι. Η τροπολογία 72 της κυρίας Μπόσκουρτ ε, γράφει ότι δεν είμαι υπέρ, αλλά στην πραγματικότητα είμαι υπέρ. Είσαστε υπέρ του του μείον που υπάρχει στον κατάλογο. Όχι, λέει η κυρία Πάκ. Τροπολογία συμβασμού 1. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 21. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 30 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 35 με χωριστή ψηφοφορία. Τμήμα 1. Κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά θα ελέγξουμε. Πέρας. Παρακαλώ. Κατά. Καταγράφει την ψήφο σα κατά. Βγάλετε την American Express παρακαλώ από, το, από τη σχισμή λέει ο πρόεδρος και βάλετε την κάρτα ψηφοφορίας. «22 με 16 κατά γίνεται δεκτή». Δεν Γίνεται δεκτό το δεύτερο μέρος. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 38 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική, παρακαλώ. Δεύτερο τμήμα έλεγχος, ηλεκτρονικός. Πέρας. 22 με 20 γίνεται δεκτό το δεύτερο τμήμα. 23-20. Συμβαστή 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ 46, υπέρ, λέει ο πρόεδρος και πάλι. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές δεχτεί. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 49 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 50 όχι όχι εκπίπτει. 52 υπέρ. 52 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 62 με προφορική τροποποίηση 2, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 64 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 65 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 70 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 71 υπέρ, κατά αποχές καρμέλεχο. έλεγχο. Πέρας 22 με 24 απορρίπτεται. 22 με 25 καλύτερα απορρίπτεται. Τροπολογία 72. Υπέρ. 72 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 10 συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή, τροπολογία 90 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 95 <clears throat> εκπίπτει. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 107 μόνο το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό 108 υπέρ κατά αποχές δεκτή 109 υπέρ κατά αποχές δεκτή 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ <clears throat> κατά αποχές απορρίπτεται 112 σε δύο τμήματα. Μάλλον το πρώτο τμήμα που να ψηφίσουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι ελέγχεται, θα, ότι εγκρίνεται, αλλά θα την ελέγξουμε. 113 παρακαλώ να ψηφίσετε. 30 με 16 εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 116 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 1 <clears throat> υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 2 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 6 υπέρ κατά αποχές. Θα ελέγξουμε για την 6. Πέρας. 27 με 21 γίνεται δεκτή. Πάμε στην 7. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 9. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 10. Υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η τελική ψηφοφορία τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Σαράντα με μία ψηφοκάτα και τρεις αποχές γίνεται δεκτή. Συγχαρητήρια στην εισηγητρία. Αν μπορούσαν οι λαοί της Βοσνίας Ερζεχοβίνης να έχουν την ίδια σύμπνοια όπως η Επιτροπή μας, θα ήταν πολύ θετικά τα πράγματα. Παρακαλώ. Σχόλιο χωρίς ε, μικρόφωνο. Είναι κέρδος και για τις δύο πλευρές, λέει ο πρόεδρος. Συγγνώμη, αλλά έτσι είναι. Αυτό είναι μη... η άποψή μου ότι καλύτερα να χάνεις φίλους παρά να χάνεις εχθρούς έτσι. Περνάμε στο Μαυροβούνιο. Ο Τσάρλ Στένοκ θέλει να πει κάτι γιατί δεν είχε δυνατότητα να λάβει το λόγο χθε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μπόρεσα να μιλήσω χθε. Θα είμαι συνοπτικότατο. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλου του σκιώδει εισηγητέ για τι επιτυχεί συνομιλίε και διαπραγματεύσει που είχαμε προκειμένου να εξεύρουμε συμβαστικέ λύσει είναι μια θετική εξέλιξη αυτή του Μαυροβουνίου ως ε, χώρα σε σχέση με τα υπόλοιπα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι υποψήφια και διπλωματεύομαστε μαζί τους, ιδίως για τα κεφάλαια 23-24, δικηστικό κλάδος, ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιοσύνη και κράτος δικαίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ε, το ξέπλυμα παράνομου χρήματος και τη συμμετοχή των γυναικών στο δημόσιο βίο, την προστασία των ε, ε, ανηλίκων και των ε, μειονοτήτων καθώς και των λαών; Είναι ένα παράδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες της γειτονιάς αυτής, της γεωγραφικής αυτής περιοχής στο Μαυροβούνιο. Απλώς πρέπει να επιληθούν κάποια συνοριακά ζητήματα με την Κροατία. Δυστυχώς βεβαίως υπήρξαν πρόσφατα επιθέσεις κατά δημοσιογράφων που πρέπει να ερευνηθούν πλήρως ώστε οι αυτούργοι να προσαχθούν ε, ενώπιν της δικαιοσύνης. Πάντως γενικώ υπάρχει συνένεση μεταξύ όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας και από τους πολίτες της χώρας ως προς τον δρόμο τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Έχουμε 130 τροπολογίες και 17 συμβαστικές. Ελπίζω η έκθεσή μου να εγκριθεί με ευρία πλειοψηφία σε αυτήν την εκτροπή. Ευχαριστώ. Έχετε σχόλια. Όχι. Προτού ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Θέλω να χαιρετήσω τον γερουσιαστή Χωσέ Πουροτόρες, ο οποίος είναι μέλος της γερουσίας του Μεξικού και τον κύριο Τόρο Γκαρίτα, που είναι γενικός γραμματέας για τα κοινοβουλευτικά θέματα της Μεξικανικής Γερουσίας. Καλώς ήλθατε και οι δύο. Μετά από την επίσκεψη του Πρόεδρου Σούλτ τον προηγούμενο Φεβρουάριο, οι σχέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Μεξικανικό Κοινοβούλιο έχουν αναβαθμιστεί <clears throat> και χαιρόμαστε πάρα πολύ μπορούμε να έχουμε αυτή την τόσο καλή συνεργασία για την βελτίωση των δεσμών μας. Σας ευχαριστώ που πήρατε το χρόνο να έρθετε να παρακολουθήσετε τις εργασίες μας. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία τη συμβαστική τροπολογία 1 στην έκθεση Τάνοκ. Ψήφι υπέρ, κατά αποχέ δεκτή. Τροπολογία 25. Τότε δεν το λέει καλά ο κατάλογος, λέει ο πρόεδρος. Συμβαστική 2. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασκή 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 42. Υπέρ κατά από χιές απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά από χιές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά εγκρίνεται. Παρακαλώ. 46 υπέρ κατά από χιές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 6 ε, λέει ο πρόεδρος 5 εννοεί Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ. 6 και πάλι υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 57 <clears throat> ψήφι υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 58 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 63 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 75 υπέρ κατά αποχές δεκτή 76 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 10 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, τροπολογία 82 υπέρ. Πού είναι 82 λέει ο πρόεδρος. 70. 87 είναι κάπως μπερδεμένος ο κατάλογος λέει ο πρόεδρος. 87 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 112 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ 115 έλεγχος λέει ο πρόεδρος προηγουμένως ηλεκτρονικός πέρας 34-17 γίνεται δεκτή. 116 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 110, 118 εκπίπτει, 119 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 14 υπέρ. <clears throat> Κατά αποχές δεκτή. 127 υπέρ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 128 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 130 υπέρ, κατά. Αποχές θα κάνουμε έλεγχο. περας πληροφορια ψηφοφορίας. 28-26 εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. απόχε δεκτή. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Σύμβασκη 16 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Προφορική τροποποίηση στην αιτιολογική σκέψη σε. Που είναι πάλι προφορικά τροποποιημένη προφορική τροπολογία αν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται, εγώ θα ψηφίσω λοιπόν. Ψήφι υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 9 ψήφι υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 10 υπέρ, <clears throat> κατά αποχές δεκτή. 11 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 17 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. 52 υπέρ, 3 ψήφοι κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Προχωρούμε τώρα στην επόμενη έκθεση του κυρίου Χάουιτ. Θέλετε να κάνετε κάποια σχόλια, κύριε Χάουιτ. Δύο από τις τροπολογίες που συζητήσαμε χθες δεν είναι σωστές στον κατάλογο ψηφοφοριών. Η πρώτη αφορά τη συμβιβαστική 13. έστειλε σχετικό email στην γραμματεία προκειμένου να διορθωθεί και να επιστρέψει στην... Μάλλον επέστρεψε η προηγούμενη εκδοχή, θα πρέπει να γίνει κάποια διαγραφή, λέγοντας ότι πρέπει οι αρχές να ε, γκρίνουν αγγίσεις για τον νόμο περί μαζικής ενημέρωσης, ώστε να συμφωνηθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις με συμφωνία της δημοσιογραφικής κοινότητας της χώρας. Αυτό για την 13 και έπειτα η προφορική τροπολογία 6. Μετά τη συζήτηση συμφωνήθηκε αυτή με παρέμβαση του κυρίου Κούκαν για το θέμα της δίγλωσης εκπαίδευσης. Η νέα διατύπωση εδώ θα λέει τονίζει ταυτόχρονα την σημασία της πρόθεσης χωρίς να είναι υποχρεωτικός ο χαρακτήρας και την δίγλωση εκπαίδευση. Τα υπόλοιπα διαγράφονται. Η μόνη αναφορά στη δίγλωση εκπαίδευση είναι η σημασία της προώθησης σε μη υποχρεωτική βάση την δίγλωση, της δίγλωσης εκπαίδευσης. Τα συμφωνήσαμε και με την κυρία Κονέλη, να ελπίζω να συμφωνήσουν και οι συνάδελφοι. Ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρος. Προσπαθώ τώρα να κατανοήσω τι σημαίνουν όλα αυτά. Έχουμε προφορικές τροποποιήσεις, σε προφορικές τροπολογίες, σε τροπολογίες συμβιβασμού. Είναι κάπως δυσνόητο. Συμβαστική 1. Ψηφί πέρα. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 10 υπέρ. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφεται Συμβαστική 2. Μα η 10 δεν έγινε δεκτή παρατηρή γραμματεία. Οπότε πάμε στην 13 και 14. 13 και 14 από κοινού. Σαλαβράκος Γιαννάκου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ <clears throat> κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ <clears throat> κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές γίνεται δεκτή. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 4 υπέρ. Έλεγχος για την 36. Είπα ότι απορρίφθηκε. Όχι, εγκρίθηκε. Έλεγχος για την 36 λέει ο πρόεδρος. Γίνεται δεκτή. 33-17. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Μια στιγμή, μια στιγμή. Λέει η γραμματεία. Η 22 έχει γίνει δεκτή, επομένω η συμβιβαστική 4 εκπίπτει, λέει ο πρόεδρο. Επειδή είναι δεκτή η τροπολογία 22. Πάμε στην τροπολογία 38 λοιπόν. 38. Α, πρέπει να τις ψηφίσουμε όλες 37 ψήφι υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 44 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 45 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 60 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 38 υπέρ, <clears throat> κατά αποχές δεκτή. 39 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Σύμβαστη 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και περνάμε τώρα στην 53. Ε, 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Προφορική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας. 34-23 εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 68 υπέρ. Κύριε Κορνέλσεν, παρακαλώ. Ίσως να σας παρακαλούσα να ελέγξουμε την 53. Δεν, διότι δεν είδα τους σοσιαλίστες και δημοκράτες να ψηφίζουν sorry. Πέρασε πολύ καιρό από τότε. Με συγχωρείτε. Ήταν ελεύθερη η ψηφοφορία για τους σοσιαλιστές, αλλά εάν ψήφισαν όπως εσείς, κερδίσατε. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Με συγχωρείτε, Ανδρέ. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 79 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 85 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 86 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 87 υπέρ υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή, Τροπολογία προφορική 6 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 13. Όχι, όχι, στην 95. 95 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 97 υπέρ. Κατά αποχές Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται λόγω ισοψηφία. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ναι, η προφορική τροπολογία ήταν μαζί. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται. 107 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 108 υπέρ έλεγχος για την 107. Πέρας ψηφοφορίας. 36-21 εγκρινεται Κρίμα που ο εισηγητής δεν, δεν έχει εμπιστοσύνη στον πρόεδρο, λέει ο κύριος Μπρόκ. Τον 8 υπέρ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 κατά αποχές δεκτή 122 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 127 υπέρ κατά από υπέρ και πάλι κατά αποχές δεκτή 128 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 133 υπέρ Εκατόν μάλλον υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 131 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 132 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 133 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, προφορική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, προφορική τροπολογία 4. Έλεγχος. Πέρας. 30-23 εγκρίνεται. 139 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 140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 κατά αποχές εγκρίνεται 147 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 148 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 149 υπέρ, κατά αποχές πάλι 149 υπέρ, λέει ο πρόεδρος, κατά αποχές απορρίπτεται. Παρακαλώ να συμμετέχετε στην ψηφοφορία. 150 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 151 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτει. 153 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 154 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 155 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 156 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 157 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 158 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 160 υπέρ κατά αποχές δεκτή 161 υπέρ κατά αποχές δεκτή 162 υπέρ κατά αποχές δεκτή 163 υπέρ κατά αποχές δεκτή 164 υπέρ κατά αποχές δεκτή 165 υπέρ κατά αποχές δεκτή 166 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 167 υπέρ κατά απορρίπτεται. 168 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 170 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 έλεγχος για την 6 ηλεκτρονικός έλεγχος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία 48 με 4 ψήφους κατά και 6 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Έκθεση Άννα Άννα θες να πεις κάτι. Όχι. Σύμβαση 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ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 εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κα, ναι, εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος. Πέρα της προφορίας. 20 με 35. Δεν εγκρίνεται. Αυτή ήταν η 50. 51 λοιπόν τώρα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Οι φιλελεύθεροι ψηφίζουν υπέρ κατά. Εγκρίνεται τότε. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται με το ίδιο αποτέλεσμα. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 συμβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 59 υπέρ. Κατά αποχές <clears throat> εγκρίνεται. 61 όχι εκπίτη. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 68. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 69. Υπέρ. 69. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 70. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 71. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ Δυστυχώ δεν μπορώ να, να δω τον κύριο Μπουτικόφερ. 76 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 με προφορική τροποποίηση ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 85 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 4 με προφορική τροποποίηση του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 52-1 με δύο αποχές γίνεται δεκτή συγχαρητήρια στην Άννα. Ερχόμαστε στο σχέδιο σύστασης. Μία ψηφοφορία μοναχα ηλεκτρονική, άρχιτη ψηφοφορία. Ναι, ναι. 53 με μία ψήφο κατά γίνεται δεκτή η ψήσταση. Συγχαρητήρια. Ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της σημερινής της διάταξης. Αποφασίστηκε την Πέμπτη από τη Συνέλευση των Προέδρων ότι βάσει τις διαδικασίες του άρθρου 50 με τη γνωστή διαδικασία αντιπαράθεσης θα ακολουθεί αυτή η διαδικασία. Ξέρω τι λέει το άρθρο 50 και γι' αυτό σας προτείνω να αναβάλουμε την ψηφοφορία για το επόμενο θέμα για την ε, <clears throat> έκθεση Zone για τη Δευτέρα. Εάν λοιπόν συμφωνείτε, θα ψηφίσουμε τη Δευτέρα έχοντας διαβάσει το, το κείμενο ώστε να ελέγξει ο εισηγητής ότι δεν ε, αντιβαίνει σε αυτά που έχουμε ήδη ψηφίσει. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 17. Η έκθεση Κόβαλ αλλά έχει αλλάξει η κατάσταση εδώ, γιατί έχει παραταθεί η πρόθεσμη για τις τροπολογίες και θα εκπνεύσει μετά από την επίσκεψη στο Κίεβο. Πότε λοιπόν είναι η τελική ψηφοφορία για τις τροπολογίες. 6 Φεβρουαρίου. Και η ψηφοφορία θα γίνει στις 3 Μαρτίου, λέει ο πρόεδρος. Αλλά έχω κάποιες ε, ε, σκέψεις γιατί θα έπρεπε να έχουμε πιο νωρίς την ψηφοφορία. Ίσως ε, θα έχουμε ή αλλιώς πρέπει να κάνουμε αργότερα την ε, προθεσμία για τις τροπολογίες, λέει ο πρόεδρος.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 όχι στις 6 Φεβρουαρίου να είναι προθεσμία, αλλά στις 10 ή 12 Φεβρουαρίου. Πρέπει να είναι δυνατόν να γίνουν οι μεταφράσεις μέσα σε δύο εβδομάδες. I, think if... the uh, rapporteur. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Έχουμε την κατάσταση αυτή στην Ουκρανία και στις γειτονικέ χώρε που αλλάζει κάθε μέρα. Αν πρέπει να καταδεθούν οι τροπολογίες πάνω από τρεις εβδομάδε πριν από την ψηφοφορία, αυτό είναι πρόβλημα με μια τόσο ρευστή κατάσταση. Γι' αυτό πιστεύω ότι η μετάφραση πρέπει να γίνει σε δύο εβδομάδε και όχι σε τρει εβδομάδε. φυσιολογικά είναι εντάξει, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να γίνει προβληματικό. Λοιπόν, μια εβδομάδα αργότερα από τις 6 Φεβρουαρίου, δεν ξέρω ακριβώς πότε. Συμφωνείτε? Έντεκα ή δώδεκα. Τι μέρα είναι η δωδεκα τι μερα ειναι η 11η? 11 Φεβρουαρίου, λέει ο πρόεδρος, στι 12 το μεσημέρι. Εντάξει. Κύριε Κόβαλ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, από ό,τι κατάλαβα, η κατάσταση έχει διαμορφωθεί ως Έχουμε νέα προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 11 Φεβρουαρίου το μεσημέρι. Πράγμα που σημαίνει ότι οι τροπολογίες μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλλονται και η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει στις 3 Μαρτίου. Ως τώρα έχουμε λάβει 231 τροπολογίες, πράγμα που σημαίνει ότι ήδη υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έκθεση αυτή. Θα σχολιάσω τα σχετικά ζητήματα εντό ολίγου. Ήμασταν προετοιμασμένοι για σήμερα βέβαια, αλλά το να μετακινηθεί η προθεσμία μετά την επίσκεψη της αντιπροσωπής μας στην Ουκρανία έχει νομίζω νόημα. Ε, είναι λογικό. Να ευχαριστήσω πάντως όλους τους συναδέλφους για τη δουλειά τους, να ευχαριστήσω για όλες τις τροπολογίες. Φαντάζομαι ότι θα λάβουμε και περισσότερες και θα αναζητήσουμε φυσικά και συμβαστικές λύσεις. Λίγα μόνο σχόλια από την πλευρά μου, διότι την έκθεση αυτή θα την ξαναδούμε ούτως ή άλλως φαντάζομαι αφού επιστρέψουμε από την Ουκρανία. Πρώτα απ' όλα έχω το εξή αίτημα να σας υποβάλω. Μην ε, δείτε την έκθεση αυτή σαν είναι μια έκθεση αποκλειστικά και μόνο για την Ουκρανία. Είναι μια έκθεση για το μέλλον της ανατολικής γειτονίας. Βεβαίως, το θέμα της Ουκρανίας μας απασχολεί ιδιαίτερως, θα πρέπει να βρούμε κάποιες συστάσεις, κάποιες διατυπώσεις, αλλά παρακαλώ τους και οδηγητές να μην μετατρέψουν την έκθεση αυτή σε μια έκθεση που να αφορά αποκλειστικά και μόνο το θέμα της Ουκρανίας. Στόχος της είναι να ετοιμάσουμε το μέλλον, να προλιάνουμε το έδαφος για την ε, μελλοντική εξέλιξη της σχέσης ανατολικής γειτονίας. Και θέλουμε να υπάρξει ένα πολιτικό όραμα το οποίο να εκφραστεί ξεκάθαρα και σε σχέση με τις πρόσφατες εμπειρίες μας, τα όσα συνέβησαν τον Δεκέμβριο. Σε δεύτερη φάση, ήθελα να απευθύνω και πάλι έκκληση, έκκληση προς όλους σας. Εάν μπορείτε, μην υποβάλλετε τροπολογίες που να έχουν να κάνουν με ιδιαίτερα ε, συμφέροντα συγκεκριμένων χωρών. Έχουμε μόνιμες εκθέσεις πρόοδου για κάθε χώρα της Ανατολικής Γειτονίας. Έχουμε τις εκθέσεις Άριους Βόλσκι και Πετσέλ πρόσφατα για τις οποίες μπορείτε να υποβάλλετε συγκεκριμένες τροπολογίες. Μην ε, αλλοιώσουμε τώρα το χαρακτήρα της έκθεσης αυτής. Φυσικά και τροπολογίες μπορεί να είναι αιτιολογημένε, να δικαιολογούνται αλλά να προσέξουμε μην, να μην γίνει η έκθεση αυτή μια έκθεση για τον Αγκόρνο Καραμπάχ λόγω χάρη. από την ίδια την δομή του εγγράφου, ελοχεύει ο κίνδυνος αυτός, αλλά βλέπω να σειραίουν τροπολογίες που εκφράζουν διαφορετικές τοποθετήσεις και λαμβάνουν διαφορετικές θέσεις σε σχέση με τη σύραξη στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Δεν θέλω λοιπόν τέτοιου είδους τροπολογίες. Θα υπάρξει και άλλη συνάντηση βεβαίως με τους κοιόδης εισηγητές προκειμένου να καταλάβουμε τι ακριβώς θα κάνουμε σε την επόμενη φάση. Πάντως, σε θέματα εχθροπραξιών, υπαγωμένων ε, εχθροπραξιών ε, σειράξεων, θα πρέπει να προσέξουμε τι πολιτικό ρόλο θέλουμε να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα και να μην επικεντρωθούμε στο ποιος έχει περισσότερο δίκιο από τον άλλο σε μια σύραξη, σε μια σύγκρουση. Αυτό είναι σφάλμα. Η πλειονότητα πάντως των τροπολογιών συμβάλλουν στη βελτίωση της έκθεσης. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους συναδέλφους, ιδίως για τις τροπολογίες που μας θυμίζουν ότι Ακόμη και σήμερα οι χώρες της ανατολικής γειτονίας φαίνεται να βρισκόνται σε δυσκολότερες πολιτικές συνθήκες από ό,τι περιμέναμε ή επίσης δεν υπεγράφει η συμφωνία συμφωνια σχέσης με την Ουκρανία Παρόλα αυτά έχουν σημασία οι σχέσεις με τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας και οι πόρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πύλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανοιχτές για αυτές. Ευχαριστώ λοιπόν όλους για τις τροπολογίες τους, ιδίω για όσους καλούν για την απελευθέρωση των καθετών θεωρήσεων. Και για τις ε, ε, ευκαιρίες σε σχέση με την ενεργειακή μας πολιτική. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Mr. Mr. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κόβαλτ. Τώρα το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές. Και με μεγάλη τιμή δίνω το λόγο στον εαυτό μου, λέει ο Προεδρεύων, που είμαι σκιώδης εκ μέρους του ΕΛΚ. Η έκθεση αυτή φτάνει σε δύσκολες στιγμές για τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Συμφωνώ με αυτό που λέτε ότι δεν πρέπει την έκθεση αυτή να την χρησιμοποιούμε για τα συμφέροντα της μια ή της άλλης χώρας, αλλά αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία, χτες το βράδυ για παράδειγμα στο Κίεβο, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Και πρέπει να εκφράσουμε βέβαια την ανησυχία μας για την αυξανόμενη βία στην χώρα αυτή. Συμφωνώ πάντως ότι πρέπει να περιμένουμε την ε, επιστροφή της αντιπροσωπείας από την Ουκρανία για να προχωρήσουμε. Αυτό που έχω εγώ πάντως σαν θέματα είναι ότι η αντιπροσωπεία του Αζερβαϊτζάν αποφάσισε να φύγει από το Euronest. Κάτι που είναι βέβαια κρίμα και ελπίζουμε να επιστρέψουν σε αυτό το φόρουμ διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης πρέπει να υπογραμμίσουμε με σαφήνεια, αλλά το λέει και ο εισηγητής, ότι καμία χώρα στην ανατολική εταιρική σχέση δεν πρέπει να χρησιμοποιεί βία ή να απειλεί άλλη χώρα για να επιλύσει διμερείς διαφορές. Ας περιμένουμε λοιπόν πόσο δύο-τρεις εβδομάδες ακόμα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στις χώρες αυτές μέχρι το Φεβρουάριο. Και σε αυτήν την θητεία του Κοινοβουλίου θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την έκθεση και ελπίζω η ανατολική εταιρική σχέση να μην υπονομευθεί από τον μεγάλο μας εταίρο στην ανατολική σχέση που είναι η Ρωσία. Ευχαριστώ. Ωραία. Φλανκενστάιν από τους σοσιαλιστές. Είναι ο σκιώδης των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ καλή η βάση που μας έχει δώσει με το εγγραφό του ο εισηγητής και υπάρχουν μονάχα μερικά σημεία τα οποία θέλω να σχολιάσω. Λέει ο εισηγητής στην αιτιολογική του έκθεση ότι ο στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε και να προαγάγουμε κοινέ αξίες. Αυτό είναι σωστό. Γι' αυτό εγώ δεν συμφωνώ ιδιαίτερα με αυτό το οποίο λέγεται στην αιτιολογική σκέψη α εδώ δίνουμε την εντύπωση ότι εμεί θέλουμε να εξαγάγουμε τις αξίες μας. Όχι, μιλάμε για κοινέ αξίες οι οποίες έχουν ήδη συμφωνηθεί στο Συμβουλίο της Ευρώπης και σε άλλα φόρα. Ένα δεύτερο θέμα που πρέπει να εξετάσουμε είναι το ζήτημα του κατά πόσο η ανατολική αυτή εταιρική σχέση συμπεριλαμβάνει αυτόματα την προοπτική μια ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα αυτός ο αυτοματισμός δεν είναι αυτόματο και στην περίπτωση του Αζερβαϊτζάν που ελπίζω ότι δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη για την ε, Euronest δεν έχουν πρόθεση να γίνουν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά θέλουν να διατηρήσουν μια στρατηγική σχέση με εμά όπως και κάνουν και για το ΝΑΤΟ. Επομένως δεν είναι για όλους η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο απότατος στόχος και αυτό θα πρέπει να το διαφοροποιήσουμε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η μόνη εναλλακτική λύση για ορισμένε χώρες της γειτονία μας. Αυτό μπορεί να μας λείπει, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Δεν είμαστε ο μόνος πόλος έλξης σε αυτή τη γειτονιά. Και γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε κανένα πρόβλημα αν επιλέγουν κάποια άλλη λύση, εφόσον αυτές οι χώρες αυτές αποφασίζουν με ελευθερία. Με ελευθερία σημαίνει χωρί την άσκηση πίεση, χωρί εκβιασμούς οικονομικούς ή στρατιωτικούς. <clears throat> Και πιστεύω ότι έχει διατυπωθεί στην τροπολογία ε, την αντίστοιχη τροπολογία το θέμα αυτό. Τέταρτο σημείο και προτελευταίο είναι προφανές ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να διαπραγματευτούμε με τη Ρωσία για την ε, συνέχεια των σχέσεων με συγκεκριμένες χώρες. Είναι ένα καθαρά ε, διμερές θέμα. Και αν θέλουμε φυσικά όποιος θέλει να προωθήσει την ειρήνη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο πρέπει να έχει επαφές και διαβουλεύσεις με τη Ρωσία και πρέπει να το κάνουμε αυτό χωρίς να δίνουμε την εντύπωση ότι κάνουμε ένα παζάρι σε βάρος τρίτων. <clears throat> και η τελευταία μου παρατήρηση Θέλω να επικυρώσω και να επιβεβαιώσω αυτά που λέει ο εισηγητής. Δεν πρόκειται μονάχα για μια εταιρική σχέση σε επίπεδο κρατικών θεσμών, αλλά πρόκειται και για την επαφή και συνεργασία των κοινωνιών των πολιτών. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από οποιαδήποτε συμφωνία ή συνθήκη μεταξύ αρχηγών κρατών ή της Κομισιόν και αρχηγών κρατών και γι' αυτό αυτό το σημείο το οποίο τόνισε ο κύριο Κόβαλ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμιστεί ακόμα περισσότερο. Χωρί την κοινωνία των πολιτών, χωρί την επαφή μεταξύ κοινωνιών των πολιτών, ημών και των γειτονικών χωρών, δεν θα μπορέσει να ευδοκιμήσει αυτή η διαδικασία. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή που έχει υπογραμμίσει λοιπόν αυτό το σημείο. Ευχαριστώ κύριε Φλέκενστάιν. Ο κύριος Βάγγελ από την ομάδα του Άλντε. Πρόεδρε, είναι εξαιρετική ιδέα, πιστεύω, η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή τροπολογιών. Οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα είναι πάρα πολλές, πράγμα το οποίο δείχνει ότι το περιεχόμενο της έκθεσης είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Και μάλιστα όχι μόνο επειδή πρόκειται για χώρες οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους πολύ όσον αφορά την ευρωπαϊκή τους προοπτική και φιλοδοξίες, αλλά επιπλέον επειδή έχουμε να κάνουμε με χώρες και έθνη με διαφορετικές αξίες. Έχουμε κοινέ αξίες, αλλά υπάρχουν και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στις κοινωνίες αυτές. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην έκθεση, κάτι το οποίο ήδη γίνεται, αλλά πρέπει να το δουλέψουμε ακόμα περισσότερο προκειμένου να αποφύγουμε παραξηγήσεις και από πλευράς των εταίρων μας, των δυνητικά εταίρων μας. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε αντιπροσωπεία με επίσκεψη στην Ουκρανία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ώστε να μας βοηθήσει να επεξεργαστούμε ακόμα παρετέρω την έκθεση αυτή. Όμως, θέλω να κάνω και μια προειδοποίηση. Δηλαδή, να αποφύγουμε την κατασκευή προκαταλήψεων. Η κατάσταση στην Ουκρανία είναι ήδη περίπλοκη και μερικές φορές έχουμε την αίσθηση ότι βρίσκεται στο χείλος φοβερής καταστροφής. Δεν θέλω να αναφερθώ σε κίνδυνο εμφυλίου πολέμου, αλλά δεν είναι μακριά από μια πολύ σοβαρή κρίση. Και δεν είμαι σίγουρος στα προηγούμενα στάδια κατά πόσο είχαμε μια αρκετά ισορροπημένη προσέγγιση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τότε δηλαδή που κολλήσαμε στον τοίχο την Ουκρανική κυβέρνηση για κάποιους πολύ συγκεκριμένους λόγους και με πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να το επαναλάβουμε αυτό στο μέλλον. Πρέπει να δείξουμε το ενδιαφέρον μας για την Ουκρανία ολόκληρη με ανατολικό και δυτικό τμήμα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι προσφέρουμε σε ολόκληρη την Ουκρανία την ευρωπαϊκή προοπτική. Αλλιώς θα υπάρξουν παρεξηγήσεις που θα οδηγήσουν σε παρετέρω προβλήματα με την Ουκρανία. Όσον αφορά τώρα την έκθεση αυτή καθεαυτή, δεν μπορούμε να αποφύγουμε βέβαια να αναφερθούμε σε παγωμένες συγκρούσεις στην περιοχή. Δεν λέω ότι πρέπει να πάρουμε θέσει σχετικά με τις συγκρίσεις αυτές, συμφωνώ με τον εισηγητή, αλλά από την άλλη μεριά θέλουμε να έχει έναν ενεργό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση και να προσπαθήσει να λύσει τις, τα, τα προβλήματα αυτά, τότε πρέπει να τα αναφέρουμε, να τα εντοπίσουμε και να τα αναφέρουμε σε σχέση με τις αξίες, τις αρχές που καθοδηγούν τις δικές μας πολιτικές. Γιατί πρόκειται και για το διεθνές δίκαιο στο κάτω-κάτω. Δεν αναφέρεται αυτό ούτε δουλειά που γίνεται σε διάφορα διεθνή φόρα σχετικά με τις παγωμένες αυτές συγκρούσεις. Συνεπώς, κάνω έκκληση να εντοπίσουμε, να αναφέρουμε τις παγωμένες αυτές συγκρούσεις για να δείξουμε έτσι το ενδιαφέρον μας και τη δέσμευσή μας προκειμένου να συνεισφέρουμε στην επίλυσή τους. Κατά τα άλλα, προσβλέπω σε καλή συνεργασία με τον ε, εισηγητή, τόσο καλή όσο ήταν και μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σούλτς εκ μέρους των Πρασίνων τώρα. Είναι πολύ καλό ότι έχουμε τώρα αυτή την έκθεση σε μια κατάσταση που έχει δραματικά χαρακτηριστικά Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε βέβαια την έκθεση της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα πάει στην Ουκρανία, εφόσον μπορέσει να πάει, γιατί κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει αυτή τη δυνατότητα. Νομίζω τώρα ότι το επίκεντρο της έκθεσης αυτής θα πρέπει να είναι η Ουκρανία, διότι η κατάσταση που παρατηρείται εκεί είναι μοναδικού χαρακτήρα. Έχουμε μια συμφωνία σύνδεσης από τη μία πλευρά, η οποία όμως δεν έχει υπογραφεί λόγω αυτής της αντιπαράθεσης που έχει προχωρήσει στην Ουκρανία μέχρι της χρήση βίας και μπορεί να οδηγηθεί σε περαιτέρω κλιμάκωση. Και υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ιδιαίτερα, είναι το θέμα του κατά πόσον συνάδει η Τελωνιακή <clears throat> Ένωση με την ε, Ένωση ε, ελευθέραν συναλλαγών που συγκροτεί η Ρωσία, η οποία θέλει να φτάνει από το Βλαδιβοστόκ μέχρι την Ουκρανία. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι συμβατά αυτά τα δύο στοιχεία. Επίση, θα πρέπει να βρούμε ένα διαφορετικό σχήμα για τι σχέσει με χώρε, οι οποίε λόγω τη ρωσική πίεση και το τονίζω αυτό, χώρε όπω είναι η Αρμενία <clears throat> και η Λευκορωσία, δεν έχουν μπορέσει να συνάψουν μια συμφωνία σύνδεση. Θα πρέπει να υπάρξει μια μορφή η συνεργασίας και εταιρική σχέσης μέσα στους περιορισμούς που υπάρχουν. Ελπίζουμε ότι και η Μολδαβία και η Γεωργία θα έχουν μια αντίστοιχη αντιμετώπιση. Αυτό το οποίο λείπει από την Ευρώπη και πρέπει να εκφράσουμε τη λύπη μας, είναι η έλλειψη μιας σωστής πολιτικής επικοινωνίας, ώστε να καταλάβει και ο πληθυσμός των χωρών αυτών τι θα κερδίσει από μια, από μια συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι το οποίο είναι αυτό και κατανοητό για τους απλούς πολίτες των χωρών αυτών σε ό,τι αφορά την καθημερινή του ζωή και έχουμε όλες αυτές τις λεγόμενες παγωμένες σειράξεις οι οποίες ε, έχουν γίνει εντωμεταξύ καυτές όπως στην Υπερνηστερία ή στον Αγκόρνο Καραμπάχ θα πρέπει να υπάρξει μια πιο έντονη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε επιτύχει ιδιαίτερα αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε και σε, σε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για τα θέματα αυτά. Ο κύριος Κύρολαφ, ο οποίος είναι <clears throat> συνεισηγητής στην Euronest για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Και συμφωνώ με τους προλήσαντες. Συμφωνώ δηλαδή ότι Τώρα συζητάμε για μια σοβαρή στάση ε, σε σχέση με το μέλλον για τις σχέσεις μας με τις γείτονες χώρες. Άρα δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Είναι ορθό ο εισηγητής που μέχρι τώρα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά να αναφέρεται και σε μακροχρόνια προβλήματα. Φυσικά χρειαζόμαστε υπομονή. Από την άλλη μεριά στην Ουκρανία τα γεγονότα καμιά φορά μας ξεπερνάνε. Πρέπει όμως να προχωρούμε με σοφία προκειμένου να μην επαναλάβουμε αποτυχίες όπως είχαμε στο παρελθόν. Και συμφωνώ με τον εισηγητή ότι χρειάζεται μια προσέγγιση κομμένη και ραμμένη ε, για τον καθένα χωριστά, γιατί δεν μπορούμε τις γείτονες χώρες μας να τις βλέπουμε όλες μαζί σαν ίδιες και να έχουμε την ίδια προσέγγιση απέναντι σε όλες. Στις πολιτικές μας δεν πρέπει να δημιουργήσουμε μια κατάσταση όπου να στοχεύουμε στην απομόνωση της Ρωσίας. Φυσικά έχουμε και διμερείς σχέσεις με όλες αυτές τις χώρες και θα έπρεπε έτσι να δούμε το θέμα. Πάντως η συνολική πολιτική μας δεν πρέπει να δημιουργεί την εντύπωση ότι προσπαθούμε να απομονώσουμε τη Ρωσία. Ακόμα περισσότερο πρέπει επικοδομητικά να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με την οικονομική συνεργασία με τις χώρες του ευξενου Πόντου. Η Βουλγαρία τώρα προεδρεύει στην οργάνωση αυτή, στον οργανισμό αυτό. Άρα έτσι μπορούμε να λύσουμε θέματα περιβαλλοντικά, οικονομικά, για τις χώρες που βρίσκονται στον εύξενο πόντο και πολλές από αυτές συμμετέχουν στην Ανατολική Εταιρική Σχέση. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί τρόποι για να το πετύχουμε. Κάτι άλλο με το οποίο συμφωνούμε με τον κύριο Βαλερ και έχω μία τροπολογία προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι παγωμένες συγκρούσεις. Αν τις δούμε σαν παγωμένες, είναι αντιπαραγωγικό. Είδαμε τι έγινε με την Γεωργία. Επιπλέον, όταν υπάρχουν εντάσεις, χρησιμοποιούνται πολιτικά. Το είδαμε με τον Αγκόρνο Καραμπάχ και με την υπερδυστερία. Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, Όλες αυτές οι συγκρούσεις μπορεί να τύχουν πολιτικής εκμετάλλευσης. Αν δεν ενδιαφερθούμε μακροπρόθεσμα, θα τα βρούμε μπροστά μας. Δείτε τι γίνεται με τους Ολυμπιακούς στο Σόλτσι. Χρειαζόμαστε ασφάλεια στις γείτονες χώρες, και στη Ρωσία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τόσους αθλητές στο Σόλτσι τώρα. Μεγάλους Ολλανδούς κλπ. Άρα πρέπει να το κοιτάξουμε και αυτό. Τέλος. Είπαμε. Προσέγγιση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της κάθε χώρας. Μεν, αλλά και μια γενική προσέγγιση από την άλλη. Δεν μπορεί να μιλάμε για εδαφική ακαιρεότητα σε σχέση με μια χώρα και σε σχέση με μια άλλη να μην το αναφέρουμε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αν επιμένουμε για την αυτοκυριαρχία, ε, ναι, αλλά θα πρέπει να είναι για όλους. Να είναι επικοδομητικό. Τι θα γίνει αν η Ουκρανία, για παράδειγμα, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην Κρυμαία, ας πούμε, θέλει αυτοδιάθεση. Τι θα βγει από αυτό. Συνεπώς να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να έχουμε την ίδια προσέγγιση απέναντι σε όλες τις χώρες όσον αφορά την ακαιρεότητα, γιατί είναι και προς το δικό μας συμφέρον. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Κύριλοφ. Ο κύριος Πόσλιτο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω αυτά που είπε ο προλαλής σας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια παλιά παράδοση ενασχόλησης με την περιοχή του Καυκάσου. Βέβαια έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα όπως της Τσεσενίας που τα έχουμε αφήσει από τα μάτια μας τελείως. Τώρα επανέρχεται με δραματικό τρόπο αυτή η προβληματική με τους Ολυμπιακούς στο Σότσι. Εγώ πιστεύω ότι οι Ολυμπιακοί αυτοί αγώνες που γίνονται 150 χρόνια ακριβώς μετά την εκδίωξη του λαού των Τσερκέζων από τον Κάφκασο και θα γίνει και μία ε, μια παρέλαση στρατευμάτων με παραδοσιακές φορεσίες των στρατευμάτων που είχαν νικήσει τους Τσερκέζους και τους διασκόρπισαν σε όλη τη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα έχουν όλα αυτά. Υπάρχει αυτή η έννοια της πυρήτης αποθήκης που χρησιμοποιούσαμε στο παρελθόν για τα Βαλκάνια, αλλά <clears throat> η πραγματική παρουταποθήκη είναι ο Κάφκασος. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο συστηματικά τον Κάφκασο και στα πλαίσια της πολιτικής γειτονία. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν θέλουμε πράγματι να αντιμετωπίσουμε σε επίπεδο ουσίας την ε, πολιτική γειτονία όπως προσπαθούμε με αυτή την έκθεση, θα πρέπει και να μην με παρεξηγείτε, να μην αφήσουμε να μας αποσπάσει όλη την προσοχή μας το θέμα της Ουκρανίας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η Ουκρανία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ έντονα το θέμα της Ουκρανίας. Θα ήταν όμως και σφάλμα πιστεύω να αφήσουμε να εστιάσουμε αποκλειστικά στην διάσκεψη του Βίλνιους και την Ουκρανία και να αφήσουμε όλα τα άλλα θέματα. Έχουμε την κατάσταση με την Αρμενία που υφίσταται πίεσης από τον κύριο Πούτιν και είναι ένα εξίσου δραματικό γεγονός αυτό ο εκβιασμός που ασκήθηκε. Χαίρομαι που αναφέρθηκε το θέμα των λεγόμενων παγωμένων σειράξεων και οι Ρώσοι ακολουθούν το διέρη και βασίλευε σε αυτή την περιοχή και πάντα αναμοχλεύουν συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις που σε όλες τις περιοχές που δεν έχει υπάρξει λύση επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. Τον Αγκόρνο Καραμπάχ λοιπόν η υπερνηστερία και άλλες τέτοιες αντιπαραθέσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. Αυτό είναι πάντα και πρέπει να είναι πάντα ένα βασικό στοιχείο για την ευρωπαϊκή πολιτική στην περιοχή του Καυκάσου. Είναι θέμα βασικό και πρέπει να παραμείνει βασικό και στην έκθεσή μας για την περιοχή του Καυκάσου πέραν των θεμάτων ενεργειακής πολιτικής. Είναι κάτι λοιπόν φυσικά το οποίο έχει μεγάλες επιπτώσεις στην ενεργειακή μας πολιτική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τένοκ. Uh, thank you very much. Uh. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ήμουν εισηγητή πριν από 10 χρόνια για όλη την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία και Επιτά ήμουν εισηγητή για την ανατολική διάσταση της γειτονία. Οπότε ξέρω πολύ καλά την περιοχή αυτή. Το μοντέλο που τώρα ε, λειτουργεί δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Βλέπουμε να έχουν αλλάξει οι ισορροπίες δυνάμεων στην ανατολική διάσταση της τότε πολιτικής γειτονίας ή πολιτική μας γειτονία. Χώρες ε, όπως η Ερμενία έχουν στραφεί προς τη Ρωσία ε, και ως προς το εμπόριο και ως προς τις ενεργειακές τους ανάγκες, αλλά δεν πρέπει να τις χώρες αυτές. Πρέπει να παραμένουν ανοιχτές οι πόρτες μας σε κάθε είδους σχέσεις που μπορούμε να αναπτύξουμε, ακόμη και αν υπάρξει τελωνιακή ένωση με το Καζακστάν και τη Λευκορωσία και τη Ρωσία τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα θέμα στο Καζακστάν, το ίδιο και στο Αζερμπαϊτζάν, που δεν ξέρουμε αν θέλει να υπογράψει ούτε καν συμφωνία συνεργασίας, αλλά ούτε και να συμπεριληφθεί στην ε, Τελωνιακή Ένωση με τη Ρωσία. Ε, αν δούμε τι έγινε στο Βίλνιους ε, πρόσφατα, μπορεί να αυξηθεί ούτως ή άλλως η πίεση από τη Ρωσία για να μην υπογράψουν οι Γεωργιανοί. Πάντως σε κάθε περίπτωση πρέπει να παραμένουμε στο πλευρό μας και ένα σχόλιο για τον κύριο Κυρίλοφ και τις παγωμένες συγκρούσεις και το κατά πόσον θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και να συνάδουμε πάντοτε με το διεθνές δίκαιο ε, καθώς και την ε, πρώτη θέση που θα πρέπει να δίνεται στην αυτοδιάθεση. Κύριε Κυρίλοφ με συγχωρείτε αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Η ίδια η Δύση είναι γεμάτη αντιφάσεις από τη μια. Δεν πιστεύουμε στην ε, εδαφική παρέμβαση, επιτρέπουμε την αυτοδιάθεση, αλλά για κάποιες περιοχές όπως το Κουρδιστάν έχουμε διαφορετική στάση. Και θα μπορούσαμε να δεχτούμε την παρουσία της ε, προσωρινής κυβέρνησης του Κουρδιστάν ενώπιον της Επιτροπής μας, αλλά και με τον Μιλόσεβιτς είχαν ε, υποθεί διαφορετικά επιχειρήματα, αλλά κανείς δεν είχε συμφωνήσει λόγω χάρη με την θανάτωση Κούρδων από τον ε, Χουσέιν. Λοιπόν, η αυτοδιάθεση είναι και η είναι σίγουρα δύο σημαντικές αρχές του διεθνούς δικαίου αλλά κάθε χώρα κρίνει, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πράγματα από τη δική της σκοπιά και ανάλογα με το ευρύτερο γεωπολιτικό σκηνικό. Εγώ σέβομαι και τις δύο αρχές, αλλά το ποια θα υπερισχύει και ποια θα εφαρμόζεται ε, συστηματικά ως πρώτη προτεραιότητα είναι κάτι που δεν μπορεί πάντοτε να ισχύει. Ευχαριστούμε η κυρία Λιούτσεβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω συζητούμε μία έκθεση που στόχο είχε να εξεύρει κάποια ισορροπία και μια θετική προσέγγιση προς όλες τις χώρες της ε, περιοχής, όχι μόνο προς μία. Αυτό είναι κάτι που και ο εισηγητής και οι σκιώδεις θα πρέπει να ε, το ε, εξακολουθήσουν και γι' αυτό τους συγχαίρουμε. Ως προς, την, ως προς τις τροπολογίες θα πρέπει να επικεντρωθούμε, πιστεύω εγώ, στην Ουκρανία, μία από τις χώρες της περιοχής. Πρόσφατα επισκέφθηκα τη Γεωργία και τη Μαλταβία. Είδα ότι οι συνομιλίες μας εκεί και πάλι επικεντρώνονται στο θέμα της Ουκρανίας και το πόσο σημαντική είναι η χώρα αυτή για την όλη γεωγραφική ζώνη. Βεβαίως, η αναβολή μας σημαίνει ότι δεν υπάρχει ακόμα κάποια σαφής στρατηγική. Δεν υπάρχει σαφής προσανατολισμός για το τι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την κατάσταση. Η στάση αναμονής σημαίνει ότι δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά και δεν ξέρουμε πού ακριβώς στοχεύουμε. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ξαναδούμε πολύ καλά και τους επικοινωνιακούς μας μηχανισμούς βεβαίως. Συμφωνώ απολύτως με όσο είπε ο κύριος Φλέκενστάιν ότι δεν μπορούμε να ε, εξάγουμε αυτόματα τα μοντέλα, το δικό μας ευρωπαϊκό μοντέλο και τις δικές μας αξίες. Θέλουμε να δώσουμε μια εναλλακτική εκδοχή στις χώρες αυτές και να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις ελεύθερα, ε, να κάνουν τις επιλογές που θέλουν. Ίσως να μην ενημερώσαμε σωστά, ίσως να μην ενημερώσαμε επαρκώς τους πολιτικούς ευθύνοντες ή τους πολίτες των χωρών αυτών θα πρέπει να τους προσφέρουμε κάτι ιδιαίτερα εύληπτο και να είναι άμεσα αξιοποιήσιμο, ώστε να δουν σωστά την ευρωπαϊκή τους προοπτική για το μέλλον. Αλλά δεν μπορούμε να τους υποσχεθούμε και την συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι σε αυτή την ε, χρονική φάση δεν είναι ε, απλό αυτό. Αλλά οι ίδιοι πολίτες πρέπει να καταλάβουν τα ωφέλη από τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί προς στιγμή δεν το βλέπουν. Οπότε δύσκολο θα πετύχουμε τους στόχους που ως τώρα είχαμε θέσει. Να συγχαρώ πάντως τον εισηγητή για την ιδιαίτερη προσοχή που έδωσε στην ε, εκπαίδευση και τον πολιτισμό ως θεμέλια για τη μελλοντική ένταξη η εμπάθηση των σχέσεων με τις χώρες αυτές, να ενισχυθεί η διάσταση αυτή, κάτι που θα εξασφαλίσει και περισσότερη συμμετοχή των πολιτών. Και εν τέλει, να επαναλάβω ότι αφού το έχουμε συζητήσει επανειλημμένο, αλλά χρειάζεται ισόρροπη σχέση με τη Ρωσία. Όχι μόνο με μία ξεχωριστή περιοχή. Όχι μόνο με την περιοχή του Ευξήνου Πόντου. Ε, η στρατηγική μας για την ε, Μαύρη Θάλασσα έχει παγώσει. Δεν έχει εξελιχθεί. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε από μια νέα προοπτική τις σχέσεις μας, τις σχέσεις μας με τη Ρωσία και να έχουμε μια βιώσιμη, διορατική πρόπτικη για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η σχέση της Ανατολικής Γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε ο κύριος Λάντσμπεργκης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο λόγια για την ε, γενική σύγχυση που έχει επικρατήσει στην ε, προοπτική μας. Όταν μιλούμε για εξαγωγή των αξιών μας με αρνητικά χαρακτηριστικά, επικεντρωνόμενη τελικά σε προώθηση αξιών και μοντέλων και καταπολέμηση αντιδημοκρατικών συνιστοσών. Πράγματα που θεωρούνται αντίθετα με τις δικές μας αξίες. Τι, ποιο είναι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή. Ας το δούμε στο πλαίσιο της πρόσφατης πολιτικής μας ανατολικής γειτονίας. Ας μιλήσουμε για την Ουκρανία. Είναι προφανές ότι για τη Μόσχα είναι καλύτερα να καταστραφεί η Ουκρανία παρά να έχει μια ευρωπαϊκή προοπτική η χώρα αυτή. Υπάρχει μια ε, επίθεση προπαγανδιστική, την οποία ουσιαστικά προκαλέσαμε εμείς οι ίδιοι Ευρωπαίοι. Η... Ε, μοιάζει σαν να προσπαθήσαμε να αποπλανήσουμε ένα αφελές, μια, ένα αφελές νεαρό κορίτσι. Πώς όμως να υπερασπιστούμε τελικά την Ουκρανία έναντι της ίδιας της Ευρώπης. Έχουμε αφήσει εκτεθειμένη την Ουκρανία. Η Ρωσία έχει, δεν έχει διστάσει να έρθει αντιμέτωπη με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα ενεργικής πολιτικής, πολιτισμού και θυμίζει πολλές φορές ε, κατάλοιπα του σταλινισμού. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να σταματήσουμε να επαναλαμβάνουμε παλιά συνθήματα για εταιρικέ σχέσεις. Δεν μιλάμε εδώ για εταιρικέ σχέσεις. Μιλάμε για αντιπαράθεση. Ανοιχτή αντιπαράθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λανσμπέργκης για την αδελφοσύνη ήταν το παλιό σύνθημα, αλλά τέλος πάντων. Να δώσω το λόγο και πάλι στον εισηγητή, τον κύριο Κόβαλ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλές από τις ιδέες που ακούστηκαν θα συμπεριληφθούν ε, στην τελική εκδοχή της έκθεσης εάν υποβάλλετε τις ανάλογες τροπολογίες. Πάντως, να σας θυμίσω ξανά ότι ο τελικός στόχος της έκθεσης είναι να δώσει μια πολιτική θεώρηση για την, για την μια μελλοντική θεώρηση για την πολιτική ανατολικής γειτονίας. Να σκεφτούμε ότι τις χώρες αυτές τις θέλουμε εταίρους μας, συνεργάτες μας στην ε, περιοχή αυτή. Βεβαίως θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε και άλλε αρχέ που θα θέλαμε να γίνονται σεβαστές στις χώρες αυτές, όπως το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, την ε, αυτοδιάθεση και την ακαιρεότητα, την αδευτική ακαιρεότητα. Όμως το να επικεντρωθούμε μόνο στα γεγονότα του Βίλνιους από τα τέλη της περσινής χρονιάς ή τις δικές μας επισκέψεις στη Γεωργία και τη Μολδαβία είναι στοιχεία που πρέπει να καλυφθούν και τα δύο. Όλα τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στα συμπεράσματα της έκθεσης. Το αν θα αφιερώσουμε μια παράγραφο στην κάθε μια από τις χώρες, αυτό είναι μια επιλογή που θα καθορίσει όλο το χαρακτήρα του εγγράφου. Αλλά αν περάσουμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες για τις παγωμένες συγκρούσεις στον Κάφκασο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε σε αυτή την περίπτωση μόνο για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Για να είναι ισόρροπο το έγγραφο θα πρέπει να κάνουμε λόγο και για τα σύνορα της Γεωργίας λόγου χάρη. Οπότε, το να υποβληθούν ακόμα περισσότερες ξεχωριστέ ξεχωριστές τροπολογίες θα έχει συνέπειες για την ισορροπία της όλης έκθεσης. Νομίζω στις συζητήσει συζητήσεις με τους σκιώδεις εισηγητές θα πρέπει να, επιλέξουμε που θα δώσουμε έμφαση και που όχι να φροντίσουμε να υποβληθούν τέτοιε τροπολογίε ώστε να υπάρξει ισορροπία στο έγγραφο. Διότι το έγγραφο δεν μπορεί να διατυπώνει απλώ γενικού κανόνε και γενικόλογε αρχέ. Χρειάζεται και κάποια επιμέρου προσέγγιση, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για την κατάσταση ή την παγωμένη σύγκρουση του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Να μιλήσουμε και για ε, τι απειλέ στα σύνορα τη Γεωργία και για τη Ρωσία. Προφανώ πρέπει να δοθεί προσοχή και σε αυτό το θέμα. Αλλά το ζητούμενο είναι τι θα γίνει εάν μιλήσουμε και για έναν τρίτο εταίρο στη σχέση που με τις χώρες της ε, Ανατολικής Γειτονίας. Τότε θα πρέπει να προσθέσουμε και την Τουρκία, η οποία έχει τεράστια σημασία για την όλη περιοχή του Καυκάσου σήμερα. Μην ε, διατηρήσουμε και επαναλάβουμε επάπειρον τα μοτίβα που μας έχουν ε, μείνει ως κατάλοιπα από την Σοβιετική εποχή να σκεφτούμε και άλλες ενδεχόμενες τροπολογίες, τροπολογίες που μπορεί να αναφέρουν την Τουρκία. Με ανησυχεί λοιπόν αυτή η κατεύθυνση που μπορεί να λάβει η έκθεση, αλλά θέλω οπωσδήποτε το τελικό έγγραφο να είναι ισορροπό για να έχει την στήριξη όλων σας. Εάν οι σκιώδες εξηγητές επιμείνουν σε μια τέτοια κατεύθυνση, βεβαίως θα φροντίσω και εγώ να προσαρμόσω αναλόγως τη δική μου προσέγγιση αλλά πραγματικά είναι μία από τι τελευταίε ευκαιρίε αυτού του κοινοβουλίου, αυτή τη θητεία να έχει ένα στρατηγικό έγγραφο. Μην βρεθούμε όμω σε δύσκολη θέση, εάν είναι υπερβολικά πολλέ οι επιμέρου, οι ατομικέ τροπολογίε των συναδέλφων. Διότι μετά θα υποβληθούν ακόμη περισσότερε και καινούργιε. Και το τελευταίο μου σχόλιο. Το έγγραφο επικεντρώνεται και σε κοινωνικά ζητήματα. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να στρέψουμε περισσότερο το βλέμμα μας προς το μέλλον. Εάν ασχοληθούμε μόνο με το τι γίνεται σήμερα, όπως με την έκθεση Σάριος και στο παρελθόν, τότε κινδυνεύουμε να, μην είμαστε, να είμαστε σύντομα εκτός επικαιρότητα. Ευχαριστώ λοιπόν για την στήριξή σας και για την υποβολή των κατάλληλων τροπολογιών. Ευχαριστούμε. Κλείνει αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Και όπως είπαμε και στην αρχή έχουμε νέα προθεσμία την 10 η Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι για την κατάθεση τροπολογιών. Τώρα ένα μικρό διάλειμμα μέχρι τις 11. Τότε θα αρχίσουμε την ακρόασή μας για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο Ιράν μετά την Γενέβη. 11 ακριβώς όμως.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 Υπότιτλοι AUTHORWAVE So, colleagues, I Αγαπητοί συνάδελφοι, ας αρχίσουμε με το επόμενο θέμα που έχουμε στην σημερινή ημερήσια διάταξη, είναι η δημόσια κρόση για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο Ιράν μετά τη Γενέβη. Καλωσορίζω εδώ τους δύο προσκεκλημένους μας, όσον αφορά τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράν μετά τη Γενέβη είναι ο Βάλτερ από το Ινστιτούτο του Βερολίνου για μελέτες και τον κύριο Ρόσπεκ από το Αντίστοιχο Ινστιτούτο στη Σουηδία. Είναι περιγνώμονες όσον αφορά τη δυναμική του Ιράν και την εξωτερική πολιτική και συντάκτες διαφόρων δημοσιεύσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε να έρθετε εδώ και για τις παρουσιάσεις που θα μας κάνετε. Η σημερινή ακρόαση επικεντρώνεται σε ένα ιδιαίτερο θέμα. Την ε, διάμεση συμφωνία για τα πυρηνικά, η οποία ολοκληρώθηκε χάρη στις προσπάθειες κυρίως της Βαρόνης Άστον και αρχίζει τώρα η εφαρμογή. Χτες ακούσαμε από τον Υπουργό Ευάγγελο Βενιζέλο για την συνεργασία όσον αφορά τα θέματα αυτά Τώρα θα δούμε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στο Ιράν και τα σχετικά ζητήματα. Υπάρχουν διάφορα σενάρια. Ποια είναι αυτά και ποιο πόλο θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει καλύτερα με τους στόχους της όσον αφορά την εξωτερική της πολιτική για τη σταθερότητα και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά τα θέματα ήταν και στο κέντρο της συνάντησης που έγινε το Δεκέμβριο στο Ιράν με συμμετοχή πέντε μελών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν μια αντιπροσωπεία υπό την κυρία Κρόνμπεργκ, στην οποία θα δώσω και το λόγο σε λίγο. Προηγουμένως όμως, για πέντε λεφτά έχει το λόγο η κυρία Μουνίθ, η οποία είναι η συγγήτρια για τις συστάσεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε, και ευχαριστώ κυρίως τους προσκεκλημένους μας που ήρθαν. Θα μιλήσω ισπανικά. Υπάρχει διερμηνία, οπότε φορέστε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Πριν από 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να έχει σχέσεις, αλλά σχέσεις για κυρώσεις ουσιαστικά. Επειδή ακριβώς δεν υπήρχε διάλογος με το Ιράν κατηγορίες, καταγγελίες, αρνητικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλων ε, των θεσμικών ευρωπαϊκών οργάνων για μια περιοχή η οποία γεννά συγκρούσεις, είναι αλήθεια. Δεν χρειάζεται εδώ να αναφέρουμε όλες τις συγκρούσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και μάλιστα ανοιχτέ συγκρούσεις, συνεχιζόμενες, που εξακολουθούν να υπάρχουν στην περιοχή. Πιστεύω λοιπόν ότι οι διαπραγματεύσεις και το χθεσινό αποτέλεσμα που είχαμε όσον αφορά τα πυρηνικά στο Ιράν αποτελούν τους πυλώνες των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράν. Το άλλο θέμα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η χθεσινή συμφωνία πιστεύω ότι αποτελεί μεγάλη διπλωματική επιτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι το κύριο θέμα στο οποίο αφοσιώθηκαν οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της κυρίας Άστον. Επιτυχία για την οποία πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας, γιατί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέκρινε, επικρίνει συχνά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Θέσεων. Εδώ όμως έγινε ένα πολύ μεγάλο ιστορική σημασία βήμα, μια που αποδέχτηκε το Ιράν τις προϋποθέσεις για να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου. Γιατί από εδώ και πέρα ο εμπλουτισμός αυτός θα είναι κάτω από το ποσοστό εκείνο το οποίο απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Επιβεβαίωσε τη συμφωνία αυτή και η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας και έτσι τώρα οι επιθεωρητές της ε, οι υπηρεσίες αυτής θα μπορούν να πηγαίνουν και να ελέγχουν τις Ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Είναι λοιπόν το ελάχιστο προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί από τη δικιά της την πλευρά να άρει μέρος των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν από το 2005 μέχρι σήμερα. Υπενθυμίζω ότι το 2002 ήταν που άρχισαν διαπραγματεύσεις για συμφωνία, που όμως παρέλυσαν το 2005 ακριβώς γιατί υπήρξε το σχέδιο αυτό εμπλουτισμού ουρανίου. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια ιστορική στιγμή και από εδώ και πέρα πρέπει να οικοδομήσουμε τις σχέσεις μας με το Ιράν, να είναι επικοδομητικές, θετικές, με μια θετική προοπτική, όχι μόνο για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου ελπίζω να συνεχιστεί ο σχετικός διάλογος και τα πυρηνικά όμως από την άλλη να έχουμε διάλογο και για τα δύο αυτά θέματα γιατί ναι μεν υπήρξε απελευθέρωση κάποιων πολιτικών κρατουμένων και μάλιστα κάποιοι έχουν βραβευθεί με το βραβείο Σαχάροφ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρόλα αυτά η κατάσταση για τα ανθρωπινά δικαιώματα εξακολουθεί να είναι ανησυχητική. Τα δικαιώματα των γυναικών για παράδειγμα ή ε, άλλων ε, κατηγοριών πολιτών λεσβιών, και κλπ. Υπάρχει επίσης πρόβλημα με την ελευθερία του τύπου. Στο Ιράν το Ιούλιο πάντως έγιναν εκλογές με πολιτική αλλαγή τώρα όσον αφορά τη στάση του Ιράν απέναντι στη διεθνή κοινότητα. Ελπίζουμε να διατηρηθεί το πνεύμα αυτό και στην εσωτερική πολιτική της χώρας. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, μετά θα κάνω ενδεχομένω άλλα σχόλια αφού ακούσω τους προσκεκλημένους μας. Προς το παρόν αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει υπόψη της τα εξή. Πρώτον, την αναγκαιότητα να είναι βιώσιμο το νέο αυτό πλαίσιο σχέσεων και να υπάρξει αντιπροσωπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράν. Έτσι ώστε να υπάρχει μία δίωδος διαλόγου και με τις Ιρανικές αρχές αλλά και με όλους τους πολιτικούς παράγοντες, την κοινωνία των πολιτών εκεί κλπ. Εφόσον δεν υπάρχει δίωδος επικοινωνίας, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το πρώτο εμπόδιο, πώς να έχουμε διάλογο. Δεύτερον, όπως είπα και πριν, πρέπει να υπάρξουν με σοβαρό τρόπο σχέσεις με διάλογο όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα με αποτελέσματα όπως είχαμε και για τα πυρηνικά. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το γεγονός ότι αποτελεί δύναμη στην περιοχή το Ιράν. Το Ιράν λοιπόν πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες περιφερειακού διαλόγου και να συμμετέχει και στο διάλογο όσον αφορά τη Συρία. Και πρέπει να στηρίξουμε τα Ηνωμένα Έθνη και να μην αφήσουμε αυτοί που κρατούν σκληρή γραμμή να επιβάλλουν τη δικιά τους άποψη. Γιατί ο πιο επικοδομητικός τρόπος προκειμένου να πετύχουν οι διαδικασίες που έχουν αρχίσει είναι η συμμετοχή όλων των παραγόντων, άρα και του Ιράν που έχει μεγάλη δύναμη. Θα αναφερθούν η συγκεκριτική διάσταση επίσης να συμμετέχει, κάτι που, για το οποίο θα μας μιλήσουν και οι προσκεκλημένοι μας δίχως άλλων. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να αρχίσει επίσης διάλογος και σε άλλους τομείς. Λαθρεμπόριο ναρκωτικών, αλλά και άλλα θέματα που ενδιαφέρουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα, αλλά και το Ιράν. Αυτά ήταν τα σημεία που ήθελα να σας αναφέρω. Θα ακούσουμε τώρα τους προσκεκλημένους μας που σίγουρα θα εμπλουτίσουν με τις παρεμβάσεις τους το κείμενο το οποίο ετοιμάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κυρία Μουνής για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Η κυρία Κρόνπερκ τώρα έχει το λόγο που είναι πρόεδρος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις μας με το Ιράν. Θα μας ενημερώσει για την τέταρτη διακοινωνιστική συνάντηση που έλαβε χώρα 12 με 18 Δεκεμβρίου στο Ιράν, αν δεν απατώμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να σας ενημερώσω για το ταξίδι της αντιπροσωπείας μας στο Ιράν. Συναντήσαμε διαφορετικές ομάδες συνομιλητών, εκπροσώπους κυβέρνησης από το, από το Κοινοβούλιο του Ιράν, Κοινωνία των Πολιτών, ΜΚΟ, εκπροσώπους ε, οργανισμών του ΟΗΕ και τους πρεσβευτές των ε, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράν. Και τους δύο ε, βραβευμένους με το βραβείο Σαχάροφ στο Ιράν. Ο κοινοβουλευτικός διάλογος είναι ουσιαστικά σε εκκρεμότητα εδώ και πολλά χρόνια μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ιράν. Συναντήσαμε πολιτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο, θρησκευτικές ε, μειονότητες όπως είναι οι Εβραίοι και οι Σουνίτες, ομάδες γυναικών, τη λεγόμενη αντιπολίτευση, για μας η αντιπολίτευση που είναι περίπου 90 μέλη του Κοινοβουλίου <clears throat> στο Ιράν υποστηρίζουν την κυβέρνηση ενώ οι άλλοι 200 είναι πιο σκληροπυρηνικοί και πιο συντηρητικοί. Η συζήτησή μας με το Ιρανικό Κοινοβούλιο έλαβε χώρα σε μια Ε, στιγμή που είχε εγκριθεί από τις ΗΠΑ ένας περαιτέρω κατάλογος εταιριών από το Ιράν που θα πρέπει να τεθούν σε εμπάργο. Αυτό του δημιούργησε την εντύπωση ότι δεν μπορούν να εμπιστεύονται τις ΗΠΑ. Είπε βέβαια ο Υπουργό Εξωτερικών του ότι δεν ήταν παραβίαση της Συμφωνία της Γενέβη και αυτό θα, οι διαπραγματεύσει θα συνεχίσουν. Αυτά μας σα δείχνουν τι εντάσει που υπάρχουν μέσα στο Ιρανικό Κοινοβούλιο. Συναντήσαμε λοιπόν τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος είναι πολύ ανοιχτός για ενδεχόμενες αλλαγές στην εξωτερική πολιτική του Ιράν. <clears throat> Ενδιαφέρεται για τις καλές σχέσεις με τους γείτονές του και αντιμετώπισαμε και το θέμα της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας και των σχέσεων του Ιράν με τις χώρες αυτές. Ο Υπουργός κ. Σαρίφ υπεγράμμισε την ε, σημασία του έργου της κυρίας Άστον, είπε ότι πρέπει να την αναγνωριστεί η προσπάθειά της για τη Συρία και τις διαπραγματεύσεις. Είδαμε και τον ε, αρμόδιο υπουργό, ο οποίος ήταν πρώην υπουργός οικονομικών, για τις ε, κυρώσεις που είπε ότι αυτό οδήγησε σε μία αύξηση κατά 10 ή 20% του κόστου συναλλαγών για τις ε, εμπορικές συναλλαγές και είπε ότι οι καταναλωτές δεν προτιμούν τα κινέζικα προϊόντα, θα προτιμούσαν να έχουν ευρωπαϊκά προϊόντα στο Ιράν. Και υπάρχουν πολλές τώρα εμπορικές αποστολές οι οποίες βρίσκονται στο Ιράν. Για το θέμα του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί αυτό ήταν από τα πιο σημαντικά θέματα που μας απασχόλησε. Συναντήσαμε τους βραβευμένους με το βραβείο Σαχάροφ. Μας ζήτησαν να θέσουμε ορισμένα θέματα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κάτι το οποίο το πράξαμε. Χαρήκαν πολύ να μας συναντήσουν. Έγινε αυτή η συνάντηση σε την πρεσβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στη συνέχεια υπήρξαν πολλές συζητήσεις, ποιος ήταν υπεύθυνο για αυτή τη συζήτηση, η πιο σκληρή πτέρυγα του Κοινοβουλίου ζήτησε να μάθει από τον αρμόδιο Υπουργό και την Πρεσβεία, αλλά δεν υπήρξε κάποια ακύρωση στις επισκέψεις μας, όλα πήγανε πολύ καλά. Το μόνο αρνητικό στοιχείο ήταν ότι το σπίτι των βραβευμένων ήταν, έγινε αντικείμενο επιδρομών από ομάδες στη συνέχεια. <clears throat> Μιλήσαμε με τον κύριο Μουσάβεν και Κερούμπιαν και αναφέρονται ότι θα ξεκινήσει και η διαδικασία με τα δύο αυτά άτομα. Σε επίπεδο διαλόγου το Ιράν δεν έχει επιτρέψει την ε, πρόσβαση του ειδικού εκπροσώπου από τα Ηνωμένα Έθνη για το Ιράν. Παρ' όλα αυτά έχουν δεχτεί τον εκπρόσωπο του ΟΗΕ για τις επιτροπές για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η κύρια αυτή δεν έχει φτάσει ακόμα στο Ιράν. Ήταν όμως πολύ ενδιαφέρον το ότι <clears throat> δεχτήκανε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Συζητήσαν επίσης και το θέμα της θανατικής ποινής. Ήταν ένα από τα κύρια θέματα συζήτηση μεταξύ μας και το θέμα της θανατικής ποινή για α, αδικήματα που έχουν να κάνουν με ναρκωτικά, γιατί εκεί ε, επιβάλλονται 80% των θανατικών ποινών στο Ιράν. Συναντήσαμε τον πρώην πρόεδρο τον Αγιατολά Χραφσαζάνη και μιλήσαμε για τα θέματα της Συρίας. Είπε ότι ο λαός Συρίας θα πρέπει να καθορίσει μόνος του την τύχη του και το τρίτο τμήμα της ε, συζήτησής μας ήταν με ΜΚΟ από την κοινωνία των πολιτών. Συναντήσαμε λοιπόν τέτοιες ΜΚΟ στην ελληνική πρεσβεία και υπάρχει μια γενική εντύπωση ότι τώρα είναι πιο εύκολο να λειτουργήσουν αυτές οι ΜΚΟ στο Ιράν. Έχει προέλθει κάποια βελτίωση και οι ΜΚΟ ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένε σε σχέση με το έργο που φέρνουν σε πέρας, τους στόχους τους, την ελπίδα να έχουν εταίρους στο διεθνή χώρο. Βέβαια λόγω των κυρώσεων είχαν δυσκολίες να έρθουν σε επαφή με διεθνείς φορείς και να παίρνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό. Ασχολούνται με θέματα τοξικομανίας, ε, ε, με, με τα θέματα του AIDS, με τα θέματα των προσφύγων Υπάρχουν πολλοί πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, υπάρχουν δύο εκατομμύρια τοξικομανείς στο Ιράν. Το έργο τους λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια το πρόβλημα είναι ότι είναι υποχρεωμένοι να περνάνε από το Καζακστάν για να παίρνουν χρήματα από τους διεθνείς φορείς γιατί υπόκειται και αυτοί σε κυρώσεις. Υπήρξε λοιπόν και συμφωνία από όλους ότι ήταν απαραίτητο να υπάρξει μια εκπροσώψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράν και μιλήσαν και για τη βελτίωση των ε, ε, ανταλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο εμπορίου, περιβάλλοντος. Θα ήταν ενδιαφέρον οι Ευρωπαίους να ξέρουν περισσότερο για το Ιράν και το Ιράν να ανοίξει περισσότερο την κοινωνία του προς τον εξωκόσμο. Πολλοί από τους πρεσβευτές ήταν ιδιαίτερα ανίσχυ για τα θέματα αυτά και τη στάση την ενδεχόμενη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία που, ήταν, που θα ήταν ίσως χρήσιμα για τη στρατηγική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όχι μόνο να περιοριστούμε στα ποινικά θέματα, έχουμε πάντα τον το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέλω να αναφέρω και τρία ακόμα ζητήματα τα οποία ελπίζω θα μπορέσουν να ενταχθούν στη στρατηγική μας από την οπτική γωνία της αντιπροσωπείας μας. Πρώτα απ' όλα, <clears throat> υπάρχει μια εντύπωση ελπίδας και σπασίματος της ε, απομόνωσης αυτό. Το είδαμε μέσα στους ε, συνομιλητές μας, τους πολίτες του Ιράν, ότι περιμένουν κάποια αλλαγή. Πιστεύω ότι αν υπάρξει μια συμβολική ενέργεια όπως η δημιουργία μιας αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τεχεράνη, αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και αυτό ίσως μπορεί να ξεκινήσει με τον ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράν και να ακολουθήσει μια πλήρης αντιπροσωπεία στο Ιράν. Δεύτερον, το θέμα είναι η μείωση των εντάσεων. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι οι συζητήσεις μας, ακόμα και με τους ε, πιο σκληροπυρηνικούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους υποχρεώνουν να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό και να δουν πού θα μπορούσε να υπάρξει κάποια αλλαγή. Γι' αυτό πιστεύω ότι η διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα που πρότεινε ο Υπουργός Εξωτερικών Σαρίφ στην εκπρόσωπο Άστον στη Νέα Υόρκη θα πρέπει να προχωρήσει. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω, της, μέσω του ειδικού εκπροσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα του κ. Λαμπρινίδη να ξεκινήσει αυτό το διάλογο στο Ιράν. Ένα από τα θέματα επίσης που μας ενδιαφέρουν είναι το θέμα της ε, λαθρεμπορίας ναρκωτικών λόγω της κατάστασης στο Αφγανιστάν <clears throat> πιστεύουν ότι θα αυξηθεί σημαντικά η ροή ναρκωτικών μετά την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν και η Ευρωπαϊκή Ένωση με το, συνεργάζεται με το Ιράν, προσπαθεί να συνεργαστεί με το Ιράν σε σχέση με την επιβολή της θανατικής ποινής σε λαθρεμπόρους ή κατόχους ναρκωτικών. Θέλω να αναφέρω επίσης το ότι ο ανθρωπιστικός διάβλος που επιτρέπει τις ανταλλαγές ε, ε, φοιτητών είναι κάτι το οποίο εκτιμάται ιδιαίτερα για την δημιουργία επαφών. Θέλω να τονίσω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε επαφές για κάθε είδους ανταλλαγές με το Ιράν και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διάφορα εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προωθηθούν παραδείγματος οι πολιτιστικές ανταλλαγές οι ανταλλαγέ φοιτητών, ανταλλαγέ ε, περιβαλλοντολόγων, γιατί υπάρχουν σημαντικά προβλήματα σε τι περιπτώσει. Και από τη στιγμή που η συμφωνία της ε, <clears throat> Γενέβης πέρατωθεί, νομίζω ότι θα υπάρχουν και δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορίου με την Ευρώπη και θα πρέπει να λάβουμε και αυτές υπόψεις στα πλαίσια μια συνολική στρατηγικής. Έχουμε λοιπόν ένα παράθυρο ευκαιρία και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κρατήσει αυτό το παράθυρο ανοιχτό Σας ευχαριστούμε κυρία Κρόνμπεργκ για αυτή την λεπτομερέστατη παρουσίαση. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Πώς από το Ερευνητικό Κέντρο του Βερολίνου για 10 λεπτά. Και μετά η συνάδελφος ε, Μουνίθ θα αναλάβει την ε, προεδρία της ε, συνάντησης. Κύριε Πώς, ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Μία σύντομη για τα εσωτερικά, μία για την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και άλλη μία για την ανάγκη του να υπάρξει ευρωπαϊκή θεώρηση για τις ενδεχόμενες μελλοντικέ σχέσεις με το Ιράν. Για τα εσωτερικά της χώρας, η κυρία Κρόνμπεργκ το είπε ήδη ότι υπάρχουν ακόμη πολλές δυσκολίες, όμως το σημαντικότερο αποτέλεσμα των ε, τελευταίων προεδρικών εκλογών είναι ότι οι ομάδες που ήταν υπέρ της υπέρ ριζοσπαστικοποίησης τελικά κέρδισαν μόνο το 13% των ψηφοφόρων. Μιλάμε για εξτραμιστικές ισλαμιστικές ομάδες που ακόμη υπάρχουν, όμως η συντριπτική πλειοψηφία του Ιρανικού πληθυσμού, όπως φάνηκε από τις εκλογές, είναι υπέρ του διαλόγου και στην ίδια την Ιρανική κοινωνία, αλλά και με την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα. Η σημερινή Ιρανική κυβέρνηση ακριβώς αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα αυτό. Επίσης, αυτός είναι και αυτό είναι και το αποτέλεσμα του της ε, αποκατάστασης κάποιων εσωτερικών εντάσεων που υπήρχαν ακόμη και με τις δυνάμεις ασφαλείας αλλά και των διαπραγματεύσεων με τη διεθνή κοινότητα. Η χαλάρωση των κυρώσεων ήταν μία από τις πρώτες προτεραιότητες. Βεβαίως υπάρχει κληρονομιά ιστορική για το Ιράν από την οποία δεν μπορεί να αποσπαστεί αμέσως όμως είναι προφανές ότι ο κύριος Ρουχάνη και ο κύριος Ουμενή έχουν την ε, σωστή αντίληψη για την κατανομή των αρμοδιοτήτων. Ο κύριος Ροχάνη ε, ασχολείται με τις εξωτερικές σχέσεις, ο κύριος ε, Μοχάνη ασχολείται με, το, με τις ιδεολογικές τάσεις της κοινωνίας φρόντισε να βάλει στη θέση τους ε, την, ε, ε, τις ριζοσπαστικές εξτρεμιστικές ομάδες μιλώντας για ιδεολογικές ευελιξίες και διαλλακτικότητα. Αυτό σημαίνει ότι κατά την άποψή του το να βρεθεί μία λύση ε, δίκαιη και ως αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά δεν είναι ε, απομάκρυνση από την οδό της επανάστασης που έχει θέσει ως στόχο το Ιράν. Είναι η σημαντικότερη μάλιστα προσφορά του Χωμενή την τελευταία δεκαετία για την ε, Ισλαμιστική αυτήν δημοκρατία. Δεν παραμένει λοιπόν μόνο στη σκληρή γραμμή ερμηνεία της ιδεολογίας. Αυτό δεν είναι μια σχετική εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει ομάδα ούτε τάση εντός του, ε, του, του συστήματος εξουσίας του Ιράν να υπονομεύσει σε εσωτερικό επίπεδο ή διεθνώς α, τις λύσεις που ενδεχομένω θα εξευρεθούν. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Οι παρατηρητές τονίζουν την οικονομική κατάσταση που είναι δυσχερής και ε, προβάλλουν το επιχείρημα ότι το πρόβλημα με το Ιράν σήμερα είναι ότι έχει πέσει θύμα των κυρώσεων. Αυτό είναι μέρη αληθές κατά τα άλλα. Οι διαδικασίες διαλόγου ε, μεταξύ των Ιρανικών ελίτ είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και ο επόμενος πολύ σημαντικός λόγος είναι ότι οι ελίτ της χώρας που ασχολούνται με την ασφάλεια βλέπουν τα πρόσφατα γεγονότα στην περιοχή ως μια παρέκκληση από τις εντάσεις που έχουν υπάρξει με τη Σαουδική Αραβία κατά παράδοση και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι τα δίκτυα της Αλκάιντα ή τα μετά την Αλκάιντα δίκτυα αποτελούν απειλή όχι μόνο για την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή αλλά και για την ε, ίδια την ιστορική ασφάλεια του Ιράν. Το Ιράν έχει αρνητική εμπειρία από τον ε, Ισλαμιστικό Φονταμενταλισμό από την πλευρά των Σουνιτών και παίρνει πολύ στα σοβαρά τέτοιου είδους απειλές. Από την ε, σκοπιά λοιπόν του Ιράν υπήρξε ανέκαθεν και θα συνεχίσει να υπάρχει μια σύγκληση συμφερόντων με τη Δύση. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Ήδη το 2001 οι Δυτικοί και οι Ιρανοί αναλυτές έφτασαν στα ίδια συμπεράσματα ως προς την απειλή από τον, την τρομοκρατία η αποτίμηση αυτή από την πλευρά του Ιράν είναι σίγουρα ορθή. Εάν δούμε πώς αξιολογούν ε, οι περισσότεροι δυτικοί αναλυτές και οι δυτικοί στοχαστές και πολιτιολόγοι τα θέματα αυτά. Κοινέ απειλέ για όλους μας για πολλαπλούς λόγους. Και εδώ θα καταλήξω στη στατική θεώρηση που θέλω να αναπτύξω για την περιοχή. Ο πρώτος λόγος είναι ότι τα δίκτυα αυτά ανανεώνονται διαρχώς, αν και είναι χαλαρά και είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσει κανείς τις αλλαγές στην ηγεσία τους. Επίσης, ακόμη μπορούν να στρατολογούν και να μετακινούν τους πολεμιστές τους αλλά και τις ειδικές τους γνώσεις από την περιοχή της ε, Βορείου Αφρικής στη Συρία, στο κέρας της Αφρικής, στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν είναι ομάδες και δίκτυα που λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο και πρέπει να τους δούμε ως στρατηγικούς παράγοντες από μόνος τους. Το Ιράν και η Σαουδική Αραβία τα τελευταία 30 χρόνια έχουν ε, ανεύθυνα παίξει το χαρτί των Σιητών και των Σούνιτων για να προωθήσουν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα υπονομεύοντας την ευρύτερη ασφάλεια της όλης γεωγραφικής περιοχής. Η σημερινή μας κατάσταση δεν μπορεί να συγκριθεί με τις πικρές εμπειρίες που έζησε η όλη περιοχή τα τελευταία και τα προηγούμενα ιδίως χρόνια. Οπωσδήποτε η ε, ένταση μεταξύ Σιητών και Σουνιτών έχει ξεφύγει κάποιες φορές από τον έλεγχο και είναι πολύ δύσκολο οποιοδήποτε κράτος της περιοχής να καλύψει τις πληγές του και μόνος του να αντιμετωπίσει, μόνο του να αντιμετωπίσει αυτή, την ένταση. Αυτό μας οδηγεί στα τρία εξή συμπεράσματα. Πρώτον, δεδομένων των κοινών συμφερόντων ασφαλείας ως προς την Αλκάιντα, εμείς στη Δύση και ιδίως στην Ευρώπη θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσον θα μπορούσε να υπάρχει μια συνεργασία περί ασφάλειας ε, επικεντρωνόμενη σε αυτό το περίεργο, παράξενο και απρόσμενο στοιχείο. Μόλις το Ιράν κατανοήσει ότι δεν μπορεί να προωθήσει τα εθνικά του συμφέροντα στην ε, Ανατολική Μεσόγειο κατά και εις βάρος των δυτικών συμφερόντων, Νομίζω ότι μόλις αυτό γίνει αντιληπτό και παραμείνει σταθερό συνειδητοποίηση, τότε το Ιράν εμέσως θα παραδεχτεί ότι ε, όπως και η στρατηγική κατά παράδοση αντίστασή του κατά του Ισραήλ ήδη κατέπεσε, τότε θα καταλήξουμε στο εξής δεδομένο. Το Ιράν θα επικεντρωθεί στην οικονομία του και το Ιράν Εφόσον επικεντρωθεί στην οικονομική ανάπτυξη, στην κεντρική Ασία, στραφεί προς την κεντρική Ασία, στις καλύτερες σχέσεις με το Αφγανιστάν και άλλες χώρες, τότε το Ιράν θα μπορέσει να είναι ένας αποτελεσματικότερος εταίρος της Ευρώπης και της Δύσης. Παρά την επαναστατική του ατζέντα. Αυτά τα δύο στοιχεία συνδυαζόμενα θα μας επιτρέψουν να έχουμε μια προβλέψιμη συμπεριφορά από το Ιράν που θα συμπεριφέρεται ως κράτος έθνος ενιαίο κράτος με το οποίο θα μπορούμε να συνεργαστούμε. Έτσι λοιπόν η συνεργασία περί ασφαλείας θα μπορούσε να είναι κάτι που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Ήδη, αν δούμε τι έγινε στο Αφγανιστάν το 2001, αυτό θα μπορούσε να απασχολήσει το Ιράν για να δει γύρω του τις ε, πλέον γειτονικέ του χώρες και να φροντίσει τη γειτονιά του ίσως με κοινή αντίληψη όπως αυτή που έχει για αυτή την περιοχή η Ευρώπη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εφόσον επιληθεί ε, Εφόσον δεν επιλύεται το ζήτημα των πυρηνικών, κανένα από αυτά τα, ζητήματα, τα θέματα δεν μπορεί να προχωρήσει και να λάβει σάρκα και ουστά. Ακόμη και έτσι όμως, με, με το θέμα των πυρηνικών, το θέμα της Συρίας και τα άλλα ζητήματα της όλης περιοχής, όλα αρχίζουν να περιπλέκονται. Είναι δύσκολο μέρα με τη μέρα να τα ξεχωρίσουμε και να βρεθούν ξεχωριστές λύσεις. Πάντως, μια εταιρική σχέση μεταξύ Ευρώπης και Ιράν θα μπορούσε να ξεκινήσει μόνον εφόσον το ζήτημα των πυρηνικών ε, λάβει κάποια είδους λύση. Και οι προσπάθειες γι' αυτό έχουν ενταθεί. Η επίσκεψη ή η αποστολή ε, αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράν θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο βήμα. Ακόμη και, και μάλιστα εφόσον πετύχει ο διάλογος ε3 συν 3. Ευχαριστούμε. Πριν περάσουμε σε διάλογο με τους παρόντες εδώ, θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρούσβερ Πάρση από το Ινστιτούτο Μελετών για Ασφάλεια της Σουδίας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα συνεχίσω μετά από αυτά που είπε ο Βάλτερ, θα αρχίσω όμως από ένα διαφορετικό σημείο κίνησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το είπε και η συγγήτρια και η κυρία Κρόμπερκ επίση. Πολλά θα έπρεπε ακόμα να γίνουν όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν και να πετύχει τις προδιαγραφές τις οποίες έχει συνυπογράψει το ίδιο. Όμως είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν συμβεί και πολλά πράγματα. Και πού οφείλεται αυτό, στο γεγονό ότι στην ουσία δεν έχουμε την Ισλαμική δημοκρατία. Τουλάχιστον όχι με την πλήρη έννοια του όρου. Και χωρί τέτοιε σχέσει δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτα. Και μην ξεχνάμε ότι αν θέλουμε να φτάσουμε κάπου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, πρέπει πρώτα να έχουμε πραγματικέ σχέσει με την Ισλαμική αυτή δημοκρατία. Και σχέσει που να μην είναι απλώς η καταγγελία αυτών που δεν μας αρέσουν, αλλά πιο ουσιαστικές σχέσεις. Έτσι λοιπόν, τα διάφορα ψηφίσματα δεν έχουν αποδώσει. Χρειάζεται διάλογος και ο διάλογος είναι αμφίδρομος. Χρειάζεται λοιπόν και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ένας όρος που έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά συχνά και πιστεύω ότι είναι ορθός. Είναι σημαντικό επίσης να θυμόμαστε ότι η Ευρώπη είχε τέτοιες σχέσεις με το Ιράν παλιότερα. Είχαμε διάλογο τη δεκαετία του 90 με το Ιράν. Και στο διάλογο αυτό υπήρχαν και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εύκολα είναι να διαμαρτυρείται κανείς και να λέει ότι ο διάλογος αυτός δεν απέδωσε παρκώς, γιατί δεν έφερε όλα τα αποτελέσματα που θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση από τους εταίρους, για παράδειγμα κατάργηση της θανατικής ποινής. Είναι όμως επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι με το διάλογο αυτό οδηγηθήκαμε σε συζητήσεις και σε διαφωνίες μέσα στο Ιράν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνεπώς, όταν αρχίζει μια συζήτηση δεν σημαίνει ότι αμέσως θα έχουμε και αποτελέσματα, σημαίνει όμως ότι βάζουμε το σπόρο για να αρχίσει η συζήτηση μέσα στην ίδια την κοινωνία που μας ενδιαφέρει, κάτι το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την αλλαγή πολιτικής. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε εμείς να επιβάλλουμε στο Ιράν να κάνει αυτό που θέλουμε. Αυτό όμως που μπορούμε είναι να τους βάλουμε στο δρόμο και να οδηγηθούν εκείνοι από μόνοι τους στην αλλαγή στη συνέχεια. Όλα αυτά βέβαια είναι μέρος ενός ευρύτερου ζητήματος που είναι τελικά τι σχέσεις θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει με αυτή την Ισλαμική Δημοκρατία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι πόσο τις 100 εμπλουτισμένο ουράνιο θα έχει εδώ, εκεί, το Ιράν και μπλα μπλα μπλα. Όχι. Είναι τι σχέσεις μακροπρόθεσμα θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει με αυτή τη χώρα. Τελεία. Πρέπει λοιπόν να σχεδιάζουμε πιο στρατηγικά τις σχέσεις μας αυτές και να συζητήσουμε αν θέλουμε να έχουμε σχέσεις και τι είδους σχέσεις θέλουμε να έχουμε με αυτή τη χώρα. Πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα λειτουργεί αυτή η σχέση και τι στόχους έχει. Και δεν πρόκειται εδώ για υπογραφή ειρηνευτικών συμφωνιών ή δεν ξέρω τι από του υψηλέ τάμενου πολιτικού. Όχι, πρόκειται για τη συμμετοχή ολόκληρη τη χώρα σε μια τέτοια σχέση. Ολόκληρο του πληθυσμού. Μόνο έτσι θα αλλάξει η κατάσταση. Η πολιτική συζήτηση πολλές φορές στην Ευρώπη για το Ιράν ακούγεται σαν να έχουμε την επιλογή. Να έχουμε ή να μην έχουμε σχέσεις με το Ιράν. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να αγνοεί το Ιράν. Είναι ένα σφάλμα, στρατηγικό σφάλμα. Το Ιράν γειτονεύει με τις γείτονες χώρες μας. Και η Μέση Ανατολή είναι μια περιοχή που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Και το Ιράν είναι σημαντικός παίχτης εκεί. Συνεπώς, μετά από αυτά που είπε και η κυρία Ολμπράιτ, ο πρόεδρος των εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μια χώρα που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Και αυτό σημαίνει κάποιο κόστος, αν δηλαδή την αγνούμε αυτή τη χώρα. Και τώρα πρέπει να πληρώσουμε αυτό το κόστος. Να το ξέρουμε ότι αν την αγνοήσουμε αυτή τη χώρα θα μας κοστίσει. Σχέσεις με αυτή τη χώρα σημαίνει σκληρή δουλειά. Σημαίνει επίσης συμβιβασμούς. Συμβιβασμοί από τις δυο πλευρές εξορισμού. Και δεν πρέπει να περιμένουμε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Μακροπρόθεσμα όμως, ναι, θα πετύχουμε τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο Ιράν. Θα βοηθήσει κάτι τέτοιο και το Ιράν για να ευθυγραμμιστεί με αυτά που ζητάνε οι πολίτες του. Αλλά και γενικότερα η διεθνή κοινότητα. Συνεπώς, εδώ εμπλέκονται διάφορα ζητήματα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία για μας, όπως και για αυτούς. Ενεργειακή ασφάλεια, περιβάλλον, περιφερειακές ε, σειράξεις και καταστροφές που βλέπουμε στην περιοχή αυτή την εποχή. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα σήμερα, γιατί είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σήμερα, αλλά είναι και σημαντικά μακροπρόθεσμα, προκειμένου να μην ξαναδούμε την ίδια κατάσταση που είχαμε παλιά ξανά στην περιοχή. Συνεπώς θέλει πολλή δουλειά. Η προσωρινή συμφωνία για τα πυρηνικά είναι μια βέβαια εύθραστη. Απαιτεί πολλή βοήθεια και πολλή στήριξη από όλες τις πλευρές προκειμένου να πετύχει τελικά. Και μέρος αυτών είναι όλες οι πλευρές να βάλουν το δικό τους πετραδάκι ώστε να αλλάξει η κατάσταση και μέσα στη χώρα. Συνεπώς, είναι ζωτική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αντιπροσωπεία στην Τεχεράνη, διότι και πρακτικά διευκολύνει την κατάσταση, αλλά και συμβολισμό σημαντικός είναι. Εφόσον θέλουμε συνεργασία ή θέλουμε απλώς να καταγγέλουμε, θέλουμε διόδους, κανάλια για να μπορέσουμε να πετύχουμε την συνεργασία. Αν έχουμε μια αντιπροσωπεία επιτόπου, θα μπορέσουμε να έχουμε και τα αποτελέσματα που θέλουμε, τουλάχιστον αυτά θα είναι εφικτά. Ο Βάλτερ αναφέρθηκε στις ε, διαφορές στην περιοχή. Πρέπει να δούμε από πιο κοντά την συμφωνία αυτή για τα πυρηνικά, η οποία αποδεικνύει τι ήταν αυτό το οποίο δεν λειτουργήσε μέχρι τώρα και τι μπορεί να λειτουργήσει από εδώ και πέρα. Το τι δεν λειτουργήσε οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι αντιδρούσαν σαν να, περιμένανε να πετύχει το δικό τους το κομμάτι. Όμως δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι, διότι δεν είναι έτσι που προχωρεί η κατάσταση εκεί και οι σειράξεις. Μπορούμε να βρούμε συμμάχους, αλλά για, όταν βρίσκει κανείς συμμάχους φτιάχνει και εχθρούς. Συνεπώς, η Σαουδική Αραβία πρέπει να συμμετέχει για να λυθούν οι περιφερειακές συρρήξεις και η Σαουδική Αραβία και το Ιράν πρέπει να τα βρουν σε κάποιο επίπεδο. Και εδώ μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αλλιώ όλο αυτό το οικοδόμημα και ό,τι έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να ξεχνάει την αρχή αυτή του Zero Sum Games. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει. Πού οδηγούν όλα αυτά. Οδηγούν στο ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν με μια σειρά. Οι στόχοι όμως και οι αρχές παραμείνουν. Η πολιτική βούληση για συζητήσεις και για σχεδιασμό είναι κάτι που πρέπει να αρχίσει τώρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα διαφορετικών πραγμάτων που έχουμε μπροστά μας και μετά να καθίσουμε να σκεφτούμε τι είδους σχέσεις θέλουμε με το Ιράν. Όχι. Η συζήτηση θα κρατήσει στη συνέχεια βέβαια πολύ, αλλά πρέπει να αρχίσει τώρα. Θα πρέπει να έχει αρχίσει πριν από πάρα πολλά χρόνια. Αλλά αφού δεν άρχισε, τουλάχιστον να αρχίσει τώρα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, αρχίζει η συζήτηση. Οι συντονιστές πρώτα και μετά οποιοδήποτε άλλος θέλει να παρέμβει και να συμμετάσχει. Πρώτα εκ μέρους του ΕΛΚ, ο κύριος Αλαφράγκα, συντονιστής από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να λάβω το λόγο αργότερα, λέει ο κύριος Αλαφράγκα. Uh, Ευχαριστώ η Άννα Γκόμης από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα και πλούσια παρουσίαση που κάνατε και ο ένας και ο άλλος. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω ότι η θέση της ομάδας με όσα είπε με όσα διαπιστώσαμε από τον Νοέμβριο με την επίσκεψή μας στο Ιράν και έρχομαι τώρα από μια συνάντηση με τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Σβόποντα. Θα θυμάται και η συνάδελφος Δεκεζέρ την επίσκεψη αυτή, ότι η κρίσιμη αυτή δέσμευση, όπως ονομάστηκε, είναι πολύ σημαντική και είναι άκρος αναγκαία. Αυτό συμπέρανε και η αντιπροσωπεία μας ε, για το Ιράν, για τις σχέσεις με το Ιράν, το είπε και η ε, Τάρια. Ε, θυμάμαι τις συζητήσεις που είχαμε για τη θανατική ποινή με τόσες διαφορετικές απόψεις αλλά πραγματικά ήταν τόσο ενδιαφέρουσα η συζήτηση, ήταν τόσο μεγάλη ε, ο ζήλος όλων να συζητήσουν, να υπάρξουν ανταλλαγές απόψεων και αντιπαρα, αντιπαραβολή απόψεων, ώστε Νομίζω μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα που να είναι εύστοχα, όπως για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό που και εσείς σωστά εντοπίσατε. Το Ιράν δεν είναι αδιάφορο σε αυτά που κάνουμε, σε αυτά που λέμε. Ε, πραγματικά, όταν μιλήσαμε με τον κύριο Λαριτζάνη, ε, από την Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εντό εισαγωγικών του Κοινοβουλίου εκεί, μας είπε ότι ακριβώς λόγω της διεθνούς εκστρατείας για να σωθεί η ζωή της Σακινέα, αυτής της γυναίκας που πρόκειται να λιθοβοληθεί, προσπάθησαν, να ανέβαλαν τη δίκη και έπεισαν τη γυναίκα να δεχτεί χρήματα προκειμένου να σωθεί η ζωή της γυναίκας αυτής. Αυτό μας είπε ότι έγινε ακριβώς λόγω της διεθνούς εκστρατείας, πράγμα που δείχνει ότι ε, όντως το Ιράν νοιάζεται. Ακούει προσεκτικά και η δική μας η δέσμευση μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Αυτό για τις διμερείς σχέσεις μας και το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου. Νομίζω ότι ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι πολύ σημαντικός και για εκείνους και για μας. Και πρώτα απ' όλα το σημαντικότερο είναι ποιο του πληρώνει, ποιο του χρηματοδοτεί. Δεν γνωρίζω. Ξέρω ότι όταν πήγαμε στι Ηνωμένε μετά την επίσκεψη εκείνη με την αντιπροσωπεία τη ΑΦΕΤ, οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν αρκετή αποστασιοποίηση ως προς τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Λένε ότι δεν ξέρουν τι κάνουν στον καταβλισμό ε, Γιούρια, λόγου χάρη, όπου δεν... Ε, επιτρέπουν να υπάρχει πρόσβαση από τους απεσταλμένους της ΥΠΑ της του ΟΗΕ. Σε κάθε περίπτωση με ενδιαφέρει ποια είναι η δική σας άποψη για το Ιράν. Εάν θεωρείτε ότι το Ιράν μπορεί να είναι μια δύναμη που εάν έχει μαζί μας επικοδομητικό διάλογο μπορεί να παίξει καταλητικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Και εσείς καταλαβαίνετε όπως και εμείς ε, ότι καταλαβαίνουν μάλλον εκείνοι όπως και εμείς ότι τα συμφέροντά μας είναι κοινά όχι μόνο στην, ε, στο επίπεδο της επίλυσης συγκρούσεων ή εντάσεων στην περιοχή αλλά ακούστηκε το ζήτημα των ναρκωτικών λόγω χάρη ή ο φόβος αποσταθεροποίησης από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Αλληλένδετα αυτά τα δύο. Τι θα προκαλούσε αυτό για το Ιράν λόγω χάρη και για εκείνους και για μας. Αλλά και σε άλλους τομείς όπως η ενέργεια και όπως σωστά υπόθηκε. Και υπό αυτήν την έννοια να ρωτήσω Πώς βλέπετε το ρόλο του Ιράν ε, ως προς την Συρία. Είδαμε ότι αποσύρθη πρόσκληση για, την, ε, για τις συνομιλίες στη Γενέβη, θες μόλις, αλλά πώς πιστεύετε ότι θα αντιδράσουν. Και το δεύτερο ερώτημα είναι για τη Σαουδική Αραβία. Συμφωνώ ότι οι σχέσεις ε, Σαουδικής Αραβίας-Ιράν είναι ζωτικής σημασίας εγώ είχα την αίσθηση ότι υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο Ιράν να είναι αρμονικές οι σχέσεις από ό,τι στη Σαουδική Αραβία. Και επισκέφτηκα τη Σαουδική Αραβία μετά το Ιράν, εκεί έθεσα τα ανάλογα ερωτήματα. Αλλά πηγαίνοντας προς τη Σαουδική Αραβία και με τις ειδήσει για την γενέση συμφωνία που τώρα έχουμε, με συγχωρείτε είναι σημαντικό να το πω, υπήρχαν ε, ειδήσει και διάβασα ένα άρθρο κάπου τον έντυπο τύπο, νομίζω σε μια τουρκική εφημερίδα, ότι το Ιράν θα χρησιμοποιούσε την πυρηνική ασπίδα του Πακιστάν, που λένε ότι έχει πληρώσει η Σαουδική Αραβία, για να υπονομευτεί η ενδεχόμενη συμφωνία Ιράν και Δύσης για τα πυρηνικά. Αυτό είναι μια απέσια προοπτική. Κανείς από τους επίσημους φορείς βεβαίως δεν επανέλαβε τέτοιες κουβέντες στη Σαουδική Αραβία, όμως υπήρχε αυτή η υποψία, είχε ακουστεί και είχε γραφτεί. Μπορεί ήδη να υπήρχε ως σκέψη στα μυαλά κάποιων. Να το έχουμε και αυτό λοιπόν στα υπόψη. Τι μπορούμε να κάνουμε για να γίνει η σχέση αυτή, η σχέση Ιράν και Σαουδικής Αραβίας, διαφορετική. Και επειδή είπατε κι εσείς ότι είναι ζωτική σημασία για την πυρηνική συμφωνία και για να παραμείνει αυτή. Και τελευταίο ερώτημα. Τι γίνεται αν το Αμερικανικό Κογκρέσο μποϊκοτάρει ουσιαστικά αυτή τη συμφωνία. Τρία λεπτά κύριε παρακαλώ. Uh, uh, Θα είμαι πολύ σύντομο. Παραμένει ένα ομό καθεστώ το καθεστώ του Ιράν και το επικρίνω ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δυστυχώ έχει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα σε δημόσιε ε, θανατικές ε, ε ποινές εναντίον ομοφιλοφίλων, μπαχάι, γυναικών. Όλα αυτά είναι λοιπόν αποτροπιαστικά σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παραμένει βέβαια μια μεγάλη χώρα και μια πολύ παλιά κουλτούρα και ελπίζω κάποτε θα ξεφορτωθεί αυτή την καταστα... καταπιαστική κυβέρνηση. Αυτό το θέμα του Ιρανικού λαού. Ενδιαμέσω θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πώς. Μου λένε ότι υπάρχει μια αναδυόμενη παράξενη συμμαχία της Σαουδικής Αραβίας που ανησυχεί για την παρουσία των ΣΥΑ στην ανατολική περιοχή της Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ που και αυτό φυσικά θεωρεί ότι απειλείται μετά από τα σχόλια του Αχμάτι Νετζάντ και την προσπάθεια να αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν που ελπίζουμε ότι η διάσκεψη Γενέβης έχει αποτρέψει. Με αυτή την παράξενη λοιπόν συμμαχία που εμφανίζεται τώρα μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας. Αναρωτιέται κανείς αν όλα αυτά μπορεί να βοηθήσουν να προωθηθεί η νευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Μου είπανε ότι η Σαουδική Αραβία επειδή θέλει να έχει τώρα αυτή την καλύτερη κατανόηση με το Ισραήλ ασκεί περισσότερη πίεση μέσω του Αραβικού Συνδέσμου στην Παλαιστινιακή Αρχή για να υπάρξει κάποια συμφωνία γη εναντίον ειρήνης κτλ. Έχετε κάποιο σχόλιο σε αυτό. Βλέπετε να υπάρχει κάποια ρεαλιστική δυνατότητα να προκύψει κάτι με αυτή την παράδοξη δι... δυναμική όπου ο εχθρός του εχθρού σου γίνεται ο φίλος σου. Φαίνεται λοιπόν να υπάρχει κάποια αλήθεια ότι προωθείται μια τέτοια σύμπραξη. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια σχόλια σχετικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι έχει δημιουργηθεί ένα νέο κλίμα στο Ιράν μετά από την τελευταία διαδικασία προεδρικών εκλογών που υποστηρίζει περισσότερο το διάλογο και λιγότερο τη ριζοσπαστικοποίηση. Αλλά νομίζω ότι αυτό το κλίμα διαλόγου οφείλεται σε κάποιο βαθμό και στο καθεστώς κυρώσεων που είχε εφαρμοστεί στο Ιράν που οδήγησε σε μεγάλη λαϊκή δυσαρέσκεια <clears throat> με την κυβέρνηση. Μέσα στο πλαίσιο αυτό είναι φανερό ότι μετά από 35 χρόνια διπλωματικής απο... απομόνωσης έχουμε θετικά στοιχεία. Το Συμβούλιο Υπουργών του Ιράν είπε ότι το Ιράν έχει πράξει τα απαιτούμενα από τη δική του πλευρά για το πυρηνικό πρόγραμμα και τώρα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει το δικό της καθήκον που είναι η άρση του εμπάρκου και να μπορέσουν να απελευθερωθούν κάποια από τα 10 δισεκατομμύρια και πάνω που είναι παγωμένα τώρα στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Και οι δύο ομιλητές έχουν τονίσει ιδιαίτερα ότι μιλάμε για μια προσωρινή συμφωνία και μια πραγματική συμφωνία θα πρέπει να ακολουθήσει. Πιστεύω ότι στις σχέσεις μας με τη χώρα αυτή, που είναι φυσικά μια περιφερειακή δύναμη, που <clears throat> ανταγωνίζεται τη Σαουδική Αραβία. Θα πρέπει να σκεφτούμε όχι μόνο όλα αυτά τα θετικά στοιχεία, αλλά και τα αρνητικά. Το ερώτημά μου τώρα είναι, δεν είναι τόσο συνδεόμενο με τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι ένα ανησυχητικό στοιχείο. Πάρα πολλοί παραγνωρίζουν ότι υπήρξαν πολλές εκτελέσεις και την ε, χρονική περίοδο των ε, προεδρικών εκλογών. Θα με ενδιαφέρει όμως να ξέρω καλύτερα από την δική σας ε, άποψη πώς βλέπετε τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών στο μέλλον. Αν δεχτούν, δηλαδή αν θα δεχτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την <clears throat> προσωρινή συμφωνία και αν και οι άλλες δυνάμεις που βρίσκονται στην διαπραγματευτική αυτή διαδικασία αν το Ιράκ το Ιράν θα πρέπει όχι μόνο να περιορίσει τον εμπλουτισμό του ουρανίου στο 5% αλλά και να μειώσει την ε, ε, χρήση κεντροφύγων γιατί δεν χρειάζεται τότε αν παραμείνει ο εμπλουτισμό στο 5% μονάχα. Επομένως να περιορίσει τη δυνατότητα να αναπτύξει πυρηνική ικανότητα το Ιράν και ποια θα έπρεπε να είναι η στάση των ΗΠΑ και των άλλων δυνάμεων σε σχέση με την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ιράν τη στιγμή που παραμένει πολύς δρόμος να διατρέξουμε για τα θέματα αυτά. Δεν θα έλεγα τώρα κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο να έχουμε μια αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις φάνηκαν ότι καλύπτονται πλήρως από την ύπατη εκπρόσωπο, όπως έγινε και με τις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρξει μεγαλύτερη ελπίδα για το διάλογο. Αλλά η παρουσία του Ιράν στην ε, ε, σύραξη της Συρίας και το γεγονός ότι δεν έγινε δυνατόν να συμμετάσχει το Ιράν στη διάσκεψη Γενέβης, όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε πολύ δρόμο να καλύψουμε και πρέπει να είμαστε πιο επιφυλακτικοί σε ένα τόσο δύσκολο θέμα. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά maximum. Οι επόμενοι ομιλητέ, παρακαλώ. Η κυρία Ρομέρο. Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι στους προσκεκλημένους μας. Δεν πιστεύετε ότι κάνουμε μεγάλη χάρα στο Ιράν όταν τους βάζουμε με τους ΣΥΤΕΣ. Όταν ήταν μεγάλη αυτοκρατορία δεν ήταν ΣΥΤΕΣ. Είναι μια χώρα πολύ ενδιαφέρουσα σίγουρα το Ιράν είναι σε μια διαδικασία ανοίγματο, δεν υπάρχει αμφιβολία μετά το Αναμινετζάτ και η συμφωνία αυτή για την πυρηνική ενέργεια ακριβώς αποτελεί μέρος αυτού του σταδίου, αυτής της φάσης όπου βρίσκονται. Αλλά Νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε πολύ παραπάνω δουλειά για να υπάρξει μετάβαση στη δημοκρατία, γιατί δεν πρόκειται μόνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται και για τα πολιτικά δικαιώματα. Όταν μιλάμε για το Ιράν, πάντα μιλάμε για την κυβέρνησή του. Δεν μιλάμε ποτέ για δημοκρατική αντιπολίτευση, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο σήμερα. Οπότε η ερώτησή μου είναι, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει συμφωνία, αν σκεφτούμε και τους Σουνίτες και τους Σίτες. Γιατί μιλάμε για ένα ιστορικό, θρησκευτικό πλαίσιο, παραδοσιακό, που τελικά θέτει τις βάσεις για την εκατάσταση, ενώ πρέπει να συζητήσουμε πολιτικά. Δεν είναι σφάλμα να επιβάλλουμε αυτήν την παραδοσιακή θρησκευτική και πολιτιστική κατάσταση και όχι να προσαρμοζόμαστε στην σημερινή πραγματικότητα. Ευχαριστώ κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποια αναλλακτική λύση σε μία προσεκτική προσέγγιση με το Ιράν. Το ερώτημά μου όμως έχει περισσότερο να κάνει με την ευρύτερη περιοχή του Ιράν. Πώς βλέπετε τις σχέσεις του Ιράν <clears throat> στην ε, κατάσταση που επικρατεί τώρα στο Ιράκ. Είναι μια σχέση που έχει να κάνει με μια θέση ισχυρής χώρας έναντι ενός δορυφόρου τους. Θέλει να επιτευχθεί κάτι από την πλευρά του Ιράκ με τη σχέση αυτή με την Τεχεράνη. Και αναφερθήκατε και στον διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είχαμε στο παρελθόν με το Ιράν και τις επιπτώσεις του. Εμείς ως Κοινοβούλιο πριν από 10 χρόνια και εγώ ήμουν μέσα σε αυτή την διαδικασία, είχα αυτή την ευκαιρία να διαπιστώσω πώς υπήρξε και η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο φατριών στο Ιρανικό Κοινοβούλιο. Το ερώτημά μου είναι, καν όλα αυτά είχαν κάποιο αποτέλεσμα. Βρισκόμαστε σήμερα σε μια κατάσταση που όλοι τρέχουμε ελπίδες με τον κύριο Ροχάνη ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Αλλά δεν είμαστε ακόμα μακριά από την κατάσταση και τον πολιτικό λόγο που ίσχυε στο παρελθόν. Είπατε ότι 13% των ριζοσπαστικών ψήφισαν υπέρ του νέου Πρόεδρου. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν κάτι να κερδίσουν σε οικονομικό επίπεδο και οι οποίοι πλήττονται όταν αυξάνεται ο αριθμός των ε, εκτελέσεων. Λοιπόν, αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με εσωτερική φιλελευθερωποίηση όσο με, με σκοπιμότητα εξωτερικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Ο κύριο Μπέλντερ, ο τελευταίο μα ε, συντονιστή για το Ιράν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ και του κύριου ηγητές. Στον κύριο Πάτσι, ο οποίο αναφέρθηκε σε διάλογο Υπάρχει ιδεολογικός φονταμεταλισμός στο Ιράν που δυσκολεύει το διάλογο. Εσείς πώς κρίνετε ότι είναι εμπόδιο για το διάλογο αυτό με την Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή που θέλουμε εμεί μια διαλογικά δημοκρατική κοινωνία στο Ιράν. Αυτή είναι η ερώτησή μου και ελπίζω να με έχετε καταλάβει κατά πόσο είναι εμπόδιο στο διάλογό μας με το Ιράν αυτή, αυτός ο ιδεολογικός φωτομεταλλισμός ε, στη χώρα. Αναφερθήκατε πάντως ε, και εσείς στην διάβρωση αυτή που υπάρχει. Τώρα, ο κύριος Αλτερπόρς, εσείς αναφερθήκατε και στα προβλήματα της ε, μειοψηφίας και ανθρώπους προέλευσης Αζερμπατζάν για παράδειγμα που είναι στο Ιράν. Εσείς πώς βλέπετε την κατάσταση των μειονοτήτων στα πλαίσια της πολιτικής σκηνής έτσι όπως παρουσιάζεται αυτή σήμερα. Και από τις προσπάθειες που γίνονται μέσα στο Ιράν στην κοινωνία. Το θέμα των ναρκωτικών, για παράδειγμα, τι διάσταση έχει μέσα στην κοινωνία. Οι ακαδημαϊκές μελέτες που έχουν γίνει δείχνουν ότι και η πολιτική για τα ναρκωτικά είναι σημαντική διότι το Ιράν και ως χώρα παραγωγός αλλά και ως διακίνηση Κατά πόσο αυτό είναι εμπόδιο στην προσέγγιση της δύση με το Ιράν. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστούμε κυρία Κρόνμπερκ τώρα εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Να σχολιάσω λίγο σε αυτά που είπε ο κύριος Πάρση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μετά να ρωτήσω κάτι τον κύριο Πόστ. Πρώτα απ' όλα, αμοιβαία σεβασμό σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και στο Ιράν ακριβώ αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μα. Να μην πάμε εκεί επιβάλλοντα τι αξίε μα, αλλά να προσπαθήσουμε να υπάρχει αυτή η αμοιβαία κατανόηση και μέσω αυτή να υπάρξουν αλλαγέ. Τελικά το θέμα είναι με ποιον συζητάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πριν πάμε στο Ιράν, Είχαμε, ξέραμε ότι εκτό Ιράν υπάρχουν διάφορε οργανώσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι είχαμε συναντήσει εκτό Ιράν και τι ξανασυναντήσαμε όταν επιστρέψαμε από το Ιράν ...και αν υπάρχει feedback. Μας ε, ρωτήσαν διάφορα πράγματα πριν, εμεί πήγαμε στο Ιράν, τα ρωτήσαμε και γυρίσαμε να τους μεταφέρουμε τις απαντήσεις. Το βασικό όμως είναι ο διάλογος με τους υπεύθυνου στο Ιράν. Και το θέμα της ε, θανατικής ε, ποινή είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει πολύ σκληρή αντιμετώπιση από την κυβέρνηση. Πολλά από τα εγκλήματα όμως που τιμωρούνται έχουν να κάνουν με τα ναρκωτικά. Και εμείς βέβαια ρωτήσαμε είναι αποτελεσματική θανατική ποινή για να αντιμετωπιστεί το θέμα των ναρκωτικών. καλό θα ήταν να έχουμε κάποια στιγμή την απάντηση. Η ερώτηση μου τώρα προς τον Βάλτερ πώς. Σίτες, Σουνίτες. Αυτός ο διαχωρισμός χρησιμοποιείται πολλές φορές. Εσείς πιστεύετε ότι καλός γίνεται ή χρησιμοποιείται τελικά σε ένα παιχνίδι δυνάμεων έχει να κάνει με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, με μειονότητες, με αυτούς που είναι πιο φτωχοί ή όντω έχει να κάνει με τη θρησκεία. Δηλαδή σε αυτή την διάκριση η θρησκεία τι ρόλο παίζει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Έντς. Χέρτς. Και εγώ ως μέλος της αντιπροσωπείας για το Ιράν θέλω να πω ορισμένα πράγματα. Καταρχήν κύριε Πώς, νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε σε σχέση με, το, με τις σχέσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ιράν. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή καμία στρατηγική προσέγγιση εναντί του Ιράν. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία <clears throat> στρατηγική πέραν των επαφών της κυρίας Άστον. Τι θα πει ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ιράν, τι πρέπει να καταλάβω ότι σημαίνει αυτό το να έχουμε κάποιες επαφές, το να έχουμε εμπόριο και να δούμε αν μας αρέσει και αν μας αρέσει κάνουμε πιο στενές σχέσεις. Τι είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε. Αυτό θα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ξέρω. Και επίσης τι θα γίνει με το διάλογο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ βλέπω να το αφήνουμε αυτό κατά μέρος και να περνάμε στην έρευνα, στο εμπόριο, κοινοβουλευτικές σχέσεις κτλ. Από την άλλη πλευρά βέβαια έχετε δίκιο. Δεν μπορούμε εμείς να επιβάλλουμε στους Ιρανούς να προχωρήσουν στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει από αυτούς. Και η προσπάθεια να εξαχθούν αξίες και επαναστάσεις, αυτό δεν έχει λειτουργήσει ποτέ καλά. Για τι κυρώσει, ξέρετε ότι αυτό ήταν πάντα ένα αμφίμαχο θέμα, επίμαχο θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς ως ομάδα θεωρούμε ότι αυτό είναι τελείως λαθασμένη προσέγγιση. Είναι ήδη δύσκολο όταν δεν παίρνουν οι ο καθάλου χρήματα που θα ήθελαν να έχουν πρόσβαση σε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα χειρότερα όταν υπάρχουν μεγαλύτερες κυρώσεις. Δημιουργείται μεγαλύτερο κίνδυνο. Ποια είναι η θέση λοιπόν για το θέμα αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και εμείς μεταξύ μας. Και επίση υπάρχει μια οικονομική κρίση η οποία μπορεί και αυτή να είναι χρήσιμη για να διατηρήσει την εξουσία της κυβέρνησης εκεί. Ένα τρίτο θέμα με ενδιαφέρει το θέμα του Αφγανιστάν. Μήπως θα πρέπει να σταθούμε στο θέμα αυτό και στο θέμα της συνεργασίας <clears throat> με την ε, αντιπροσωπεία που είναι αρμόδια για το Αφγανιστάν. Τι θα γίνει με αυτά που θα γίνει το 2014 τι θα γίνει όταν αποχωρήσουν οι Αμερικανοί από το Αφγανιστάν. Μπορεί να υπάρξει λοιπόν ένα θέμα για την επιρροή του Ιράν στην περιφερειακή αυτή περιοχή χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το Αφγανιστάν και τους φόβους οι οποίοι μπορούν να προκληθούν τη ροή ναρκωτικών και την ενδεχόμενη ροή πάρα πολλών προσφύγων <clears throat> από το Αφγανιστάν. Όλα αυτά λοιπόν πιστεύω να τα αντιμετωπίσει κανείς από κοινού. Ευχαριστώ κύριε Ντουρό. Τέλος. Και μετά θα δώσουμε το λόγο πάλι. Μάλλον δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Σχέσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις των προσκεκλημένων. Συμμετέχω στη... Συμμετείχα και εγώ στην αντιπροσωπεία που πήγε στο Ιράν το Δεκέμβριο και σας άκουσα. Ξέρω και εμείς τι είδαμε επί τόπου Δηλαδή πόσο περίπλοκες είναι οι σχέσεις, ο σχετισμός δυνάμεων μέσα στην ίδια την ιρανική κοινωνία, το είπατε και εσείς τα πράγματα δεν είναι απλά. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν και τις εσωτερικές εντάσεις και την βούληση για διάλογο, θέλω κύριε Παρσί κυρίω να μας μιλήσετε λίγο για το χρονοδιάγραμμα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το χρονοδιάγραμμα στα πλαίσια ενός διαλόγου. Πώς το βλέπετε εσείς. Ξέροντας ότι η Γενέβη 2 θα λάβει χώρα κατά πάσα πιθανότητα χωρίς το Ιράν, δεν ξέρω και πού θα καταλήξει λαμβάνοντας υπόψη το εξάμεινο που έχει στη διάθεσή του το Ιράν για να θέσει σε εφαρμογή την πυρηνική συμφωνία, εσείς πώς βλέπετε το χρονοδιάγραμμα προκειμένου να γίνει πιο εντατικός ο διάλογος με το Ιράν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο όσο γίνεται καλύτερα, ζυγίζοντας τις εσωτερικές εντάσεις, την ε, συζήτηση, για να μην πω την απόφαση εντό εισαγωγικών, για την κατάσταση στη Σύρια και την πυρηνική συμφωνία που αποτελεί ένα βήμα βέβαια, ένα σκαλοπάτι στο όλο Και βέβαια με ενδιαφέρει και εμένα αυτό που ρώτησε η φίλη μου. Ξέχασα το όνομά της τώρα. Ναι, η Άννα Γκόμες, συγγνώμη. Για το θέμα των διαπραγματεύσεων και τις σχέσεις Ιράν-Συρίας στο σημερινό πλαίσιο της διάσκεψης, που δεν ξέρουμε βέβαια πού θα καταλήξει η απουσία του Ιράν. Ευχαριστούμε. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Σχέσεων, κύριε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση. να παρακολουθήσουμε τις σημερινές συζητήσεις. Εκτίμησε ιδιαίτερως πολλές από τις ευθύς παρατηρήσεις των δύο ομιλητών μας, αλλά και της κυρίας Κρόνπερκ που μας ενημέρωσε για την επίσκεψή της στο Ιράν τον περασμένο Δεκέμβριο. Με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιτρέψτε μου ίσως να ξεκινήσω με μια-δυο γενικές παρατηρήσεις. ως προς τους τομείς ενδεχόμενης συνεργασίας που μπορούμε να αναπτύξουμε με το Ιράν. Πολλά από ακούστηκαν αφορούν τομείς συνεργασίας όπου η ΕΕΔ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούν ως τομείς που πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω. Μάλιστα, αν κοιτάξετε στον ιστότοπο της ΕΕΔ για το Ιράν, το κεφάλαιο για το Ιράν, θα δείτε ποιους τομείς ε, έχουμε εντοπίσει, ώστε να διερευνήσουμε τις δυνατότητες συνεργασίας με το Ιράν όταν το πολιτικό κλίμα θα είναι κατάλληλο. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί τούτου. Κατά τα άλλα, όπως ε, ξέρουμε, οι λεπτομέρειες είναι πάντοτε είναι δαιμονικές. Μπορεί να προχωρήσουμε, χωρίς να υπάρχει λόγος, με βιασύνη. Αυτό να το αποφύγουμε. Καλό θα ήταν να είμαστε συνετοί, διότι τα χθεσινά γεγονότα είναι μία απτή απόδειξη αυτού που είπα. Χωρίς συγκεκριμένη ανάλυση για την ακολουθία των γεγονότων, δεν θα καταλαβαίναμε τι έγινε. Αλλά οι σχέσεις της Δύσης με το Ιράν είναι αντικείμενο της απόσυσης, της αναστολής, της πρόσκλησης στη Γενέβη ή είναι κάτι παραπάνω. Είναι πολύ ευαίσθητα ζητήματα αυτά και η μεταβατική αυτή περίοδος είναι ιδιαίτερα έφραστη ως ισορροπία. Δηλαδή από κάποιο είδους αντιπαράθεση έχουμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε ένα θετικό κλίμα και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, προσεκτικοί στο πώς προχωρούμε. Βεβαίως μπορώ να προσυπογράψω πλήρως στους ε, τομείς συνεργασίας που αναφέρθηκαν, αλλά να είμαστε συνετοί. Και όπως είπε ο κύριος Παρσί, να αναζητήσουμε περιπτώσεις όπου ωφέλη θα υπάρχουν για τις δύο πλευρές, τις καταστάσεις όπου τα συμφέροντα συγκλίνουν. Η προηγούμενη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναζητά τομείς συνεργασίας που είναι μη αμφιλεγόμενοι και δεν έχουν καθόλου πολιτικό χαρακτήρα, να βασιστεί σε αυτή την προσέγγιση είναι ένα ενδεχόμενο. Είδαμε ότι έχουμε ήδη κάποια επιρροή ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα λόγω χάρη στο Ιράν. Να, υπάρξει λοιπόν κάποιο είδους έλξη. Όχι απλώς να ακούγονται δηλώσεις που μας ικανοποιούν γιατί παραμένουμε πιστοί στις αρχές μας, αλλά αν θέλουμε να υπάρχει κάποιος, ε, κάποια επιρροή από πλευράς μας στο Ιράν, να καλύπτουμε τα ζητήματα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι παραγωγικός, να οδηγεί σε κάποιο αποτέλεσμα και να μην δημιουργούνται φραγμοί. Αυτές είναι οι γενικές παρατηρήσεις που ήθελα να κάνω. Ακούστηκαν επικριτικά σχόλια για την ε, θεώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σχέσης της με το Ιράν. Νομίζω ότι είναι ένα θεμητό ερώτημα να βλέπουμε αν υπάρχει τέτοιου είδου θεώρηση, αλλά η θεώρηση αυτή θα έχει ενδιαφέρον μόνο εφόσον δημιουργηθεί ε, ένα τέτοιο κλίμα. Δεν είναι μια απόφαση όπως ένα ζευγάρι που άντρας λέει στη γυναίκα θα σε παντρευτώ και θα κάνουμε και έξι παιδιά ε, και μπαίνει πρόγραμμα. Πρέπει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα και η θεώρηση αυτή ενδεχομένως να χρειαστεί να μεταβληθεί με τον χρόνο προσαρμοζόμενη στις εξελίξεις. Δεν θέλω να μακρηγορήσω περαιτέρω, περαιτέρω αλλά ίσως να πω ότι σε ό,τι φορά την ε, εγκατάσταση ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας στο Ιράν, σε γενικές γραμμές η Ευρωπαϊκή Ένωση φρονεί ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν δυνατότητες διπλωματικής επικοινωνίας, διάβλη διπλωματικού διαλόγου και στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναζητήσει τρόπους ώστε να καλύψει μια σχετική περιορισμένη μεν παρουσία στο, στην Τεχεράνη. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποστείλει υπευθύνους της ε, προσκεκλημένους των πρεσβειών των κρατών μελών, αλλά αυτό δεν ήταν αποδεκτό από το Ιράν. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε εάν μπορούμε να προλυάνουμε το έδαφος για να υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη στο μέλλον. Όμως, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι τελείως ε, θέμα μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφασίσει γι' αυτό. Έγινε επίσης ένα ενδιαφέρον σχόλιο για την ανάγκη και τρίτες χώρες να συμμετάσχουν εδώ. ιδίω η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του κόλπου να επαναθεωρήσουν τις σχέσεις τους με το Ιράν. Να τονίσω ότι την περασμένη εβδομάδα είπατε εκπρόσωπος ήταν στον κόλπο. Στον ε, αραβικό κόλπο. Έγιναν πολλές συζητήσεις εκεί και συζητήθηκε και η θέση των Σαουδαράβων ως προς το Ιράν και αυτήν την πρώτη μορφή συμφωνίας που εξευρέθη χάρη στο διάλογο του ε3-3. Επίσης, να σας επισημάνω το γεγονός ότι είναι πολύ σημαντικές οι ε, κατηδίαν συνομιλίες. Δηλαδή δεν ανάγκη να υπάρχουν επαφές μόνο σε κυβερνητικό ή σε διοικητικό επίπεδο. Υπάρχουν ένα σωρό εργαλεία, το Erasmus Mundus και άλλες ευκαιρίες, τα ερευνητικά προγράμματα πλαίσιο. Υπάρχουν τα εργαλεία για να εμπλέξουμε, να συμπαρασύρουμε και να κάνουμε το Ιράν να συμμετάσχει. αφού τη συνεργασία λοιπόν θα πρέπει να την διευρύνουμε την κατάλληλη χρονική στιγμή. Θα παραμείνω σε αυτά, θα είχα και πολύ περισσότερα να πω, αλλά νομίζω ότι ήδη είχατε πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να πω και εγώ δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι η κατάσταση σήμερα κιόλα και με την πρόσκληση του ΟΗΕ ε, προς το Ιράν να ε, συμμετάσχει στις συνομιλίες της Γενέβης και την αποστολή της, νομίζω ότι αυτό υπονομεύει το ρόλο του ΟΗΕ και του φιλελεύθερου πνεύματος που θέλουμε να εμπνέει και να διαπνέει την κοινωνία των πολιτών διεθνώ. Στη Γενέβη 2 έπρεπε να έχει προσκληθεί και το Ιράν και ξέρουμε ότι ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία πρέπει να ληφθεί με πολιτικά μέσα. Η Συρία και οι υπόλοιποι περιφερειακοί παράγοντες θα έπρεπε να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και εδώ συμπεριλαμβάνεται το Ιράν. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι το Ιράν προφανώς είναι κάτι παραπάνω από μια χώρα Σιητών. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένε Πολιτείε και το Ιράν πάνω απ' όλα έχουν κοινό συμφέρον ώστε να εμποδίσουν την εξάπλωση του φονταμεταλισμού και των εχθροπραξιών στην ε, Συρία και το Λίβανο και βεβαίως το Ιράν ως χώρα Σύτων είναι κατά τον, ε, της Αλκάιντα και της οποιαδήποτε μορφής βίας. Να δώσω τώρα το λόγο σε εσά. Πρώτα απ' όλα εσείς κύριε Πάρση και μετά εσείς κύριε Πώς. Σας ευχαριστώ για τα ερωτήματα λέει ο κύριο Πάρση. <clears throat> Εν συντομία θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο μπορώ. Ο σεχταρισμός, η, η σύγκρουση μεταξύ δογματικών ομάδων δεν είναι κάτι το οποίο προέρχεται από τη φύση, είναι απλώ κάτι το οποίο εκμεταλλεύονται οι πολιτικοί για δικού του πολιτικού στόχου. Βέβαια, όταν το ξεκινήσει κανεί αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να το σταματήσει, δεν μπορεί να το κλείσει. Αν μπορέσει λοιπόν να. Αν δημιουργηθεί αυτό, άμα βγει το τζιν από το μπουκάλι, δεν μπορεί να το σταματήσει ένα πολιτικό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ λιγότερο ιδεολογικό το Ιράν σε σχέση με τα θέματα αυτά έναντι τη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία έχει μια πιο μονομερή αντιμετώπιση, μια άποψη καθαρά δογματικό θρησκευτική σε σχέση με το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι γίνεται με τι κυρώσει. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να θυμόμαστε ότι αυτό το οποίο κάνει το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να παίζει ένα παιχνίδι ψευδεστήσεων που πιστεύουν ότι με τι κυρώσει μπορούν να πετύχουν τα πάντα. Το αφήγημα ότι οι κυρώσει έχουν αποφέρει καρπούς, είναι, το πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ απλουστευτική αυτή η αντιμετώπιση. Η νομοθεσία που περνά από την Γερουσία αυτή τη στιγμή δεν έχει το στόχο να επιτύχει ε, ή να λύσει όλα τα προβλήματα, απλώς να κάνει πιο δύσκολη τη θέση του Ομπάμα και πιο δύσκολο για τους Ιρανούς να πούν ότι έχουν ένα αξιόπιστο συνομιλητή όταν υπάρχει η πίεση των σκληροπυρηνικών στο Ιράν. Γιατί υπάρχει μια διαφορά μεταξύ αυτών που θέλουν οι πιο σκληροί οι Ρεπουμπλικάνοι και ο Ομπάμα στο Ηνωμένο, <clears throat> Ηνωμένες Και εδώ είναι το πρόβλημα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα αυτή γραμμιζόταν με την Αμερικανική στάση, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε δύο στάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και εμείς υποστηρίζουμε μονάχα αυτό που λέει εκτελεστική εξουσία και όχι νομοθετική εξουσία. Το πρόβλημα είναι ότι περισσότερε από τι ε, κυρώσει που εμεί έχουμε δεχτεί έρχονται από το Αμερικανικό Κογκρέσο και όχι από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Τώρα, δεν είναι οι κυρώσει που έχουν οδηγήσει σε αποτελέσματα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με μια τέτοια αντιμετώπιση, κυρίω ουσιαστικά αγνοεί τελείω την εσωτερική δυναμική τη κοινωνία του Ιράν. Αν δείτε το Ιράν τα τελευταία 30 χρόνια, όπω οποιασδήποτε κοινωνία που έχει περάσει από την επανάσταση σε μια μετα-επαναστατική φάση, βλέπετε ότι υπάρχει μια κίνηση παλινδρομική από την επαναστατική ιδεολογία στην μεταρρυθμιστική στάση. Αυτό γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό και ξεκίνησε πριν από τις κυρώσεις. Το να λέμε ότι ο Ρογάνιμι θέλει να αλλάξει τα πράγματα μονάχα επειδή έχουμε επιβάλει κυρώσεις είναι στο να αυτό <clears throat> επιβραβεύουμε και να συγχαίρουμε τους εαυτούς μας χωρίς να κατανοούμε την πραγματική κατάσταση. Τώρα, αν είναι πιο σημαντική η σχέση με τις ΗΠΑ ή με την με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι θα είναι διαφορετικά αυτά που θέλουν οι ΗΠΑ και θέλουν να πετύχουν και αυτά που έχουμε εμεί στο μυαλό μα και μπορούμε να πετύχουμε. Οι ΗΠΑ στο Ιράν έχουν μια δυσλειτουργική έλλειψη σχέση. Αυτή η συμφωνία του φέρνει σε μια λειτουργική μη σχέση. Πολλοί στο Ιράν θα θέλαν να έχουν μια λειτουργική σχέση με τι ΗΠΑ. Αυτό όμω είναι ακόμα μακριά, πέραν του οριζόντα. Εμείς μπορούμε να έχουμε όμως μια λειτουργική σχέση με το Ιράν πολύ καλύτερα από ό,τι μπορεί να, έχει, να έχουν οι ΗΠΑ, αν το θέλαμε και απέξουμε σωστά τα χαρτιά μας. Τελικά σε τι θα καταλήξουν όλα αυτά τα πράγματα. Και πάλι πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει μια συμφωνία που το Ιράν θα, θα απορρίψει την ε, τον εμπλουτισμό ουρανίου. Και αυτό το έχει κατανοήσει η Αμερικανική κυβέρνηση. Κάποια μορφή εμπλουτισμού ουρανίου θα γίνει στο Ιράν. Δεν μπορεί καμία συμφωνία να το εμποδίσει αυτό. Μόνο με πόλεμο μπορεί να το εμποδίσει κανείς. Αλλά πρέπει να βρείτε μετά του στρατιώτε και τα χρήματα για να το κάνει αυτό. Και αυτό δεν το έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Ομπάμα, ούτε ενδιαφέρεται για να κάνει κάτι τέτοιο. Οι μόνοι οι οποίοι υποστηρίζουν μια τέτοια στάση είναι το Κογκρέσο των ΗΠΑ, αλλά φυσικά δεν είναι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την έναξη ενό πολέμου από ΗΠΑ τι θα σημαίνει μια ομαλή και φυσιολογική σχέση με το Ιράν. Θα ήταν σαν οποιαδήποτε άλλη σχέση με μια άλλη χώρα. Θα σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να συζητάμε τα σημεία στα οποία διαφωνούμε και να υπάρχει σε καθημερινό επίπεδο αλληλεπίδραση για θέματα τα οποία δεν απαιτούν πολιτική ε, συζήτηση, είτε είναι φοιτητικέ ε, ανταλλαγέ ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που λέμε λοιπόν μια ομαλοποίηση, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ο μακροχρόνιος στόχος. Αλλά για, για το σημερινό επίπεδο δεν πρέπει απλώς να επαναφέρουμε όλα τα σημεία ε, που έχουμε με το Ιράν, να τα θέτουμε επιτάπτως και μετά να απογοητευόμαστε όταν δεν προχωράει τίποτα. Αυτό συμβαίνει πάντα, είτε μεταξύ ατόμων είτε μεταξύ κρατών δεν μπορεί να λειτουργήσει μια τέτοια στρατηγική. <clears throat> για το αν το Ιράν έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση το ότι είναι το κράτος, τι σημαίνει κράτος, ή αν είναι τέτοια θεοκρατία που να είναι πολύ μακριά από όλα αυτά που έχουμε στη Δύση. Εγώ δεν διαφωνώ απόλυτα. Αν θέλετε το Ιράν και να φύγετε από την ιδέα του hijab και του τουρμπανιού, θα δείτε ότι είναι ένα πραγματικά σύγχρονο και εξυγχρονισμένο κράτος. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι σαν και εμάς ή να βλέπουν τα πράγματα μόνο με το δικό μας τρόπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις το κάνουν. Αλλά αυτό καθε αυτό δεν πρέπει να είναι το κριτήριο για την αλληλεπίδραση με το Ιράν. Αν μιλάτε μόνο με αυτού οι οποίοι μοιάζουν σε εμά και μιλά σαν και εμά, τότε ο κόσμο μα θα γίνει πάρα πολύ μικρό. Και είναι οι συνομιλητέ μα στο Ιράν. Οι συνομιλητέ μα στο Ιράν πρέπει να είναι σε όλα τα επίπεδα. Δεν μπορεί να γίνει μια αλληλεπίδραση μονάχα σε επίπεδο Υπουργείων. Θα πρέπει να υπάρξει ένα είδο σχέσει όπου μπορεί η συζήτηση να γίνεται με ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα. Το γεγονό ότι υπάρχουν προγράμματα μελέτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν σημαίνει ότι εν καιρό αυτή η αντιμετώπιση, αυτή η γλώσσα θα μεταλαμπαδευτεί θα απλωθεί στο Ιράκ. Σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να έχουμε μια επιρροή. Και τέλος. Για να επανέλθω σε αυτά που είπε ο εκπρόσωπος της εξωτερικής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί σε κάποιο βαθμό, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τόσο καλά που έχουν φτάσει τα πράγματα να είναι, δεν θα είναι καλύτερα πολύ εύκολα. Θα πρέπει επομένως να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας και όχι να τις αποσύσουμε. Η συμφωνία αυτή και οτιδήποτε προκύψει από αυτή τη συμφωνία σημαίνει ότι πρέπει από την αρχή να δώσουμε κι εμείς κάτι. Δεν μπορούν να γίνουν τα πράγματα από μόνα τους και μετά δούμε αν θέλουμε εμείς να συμμετέχουμε σε αυτή τη συμφωνία ή όχι. Για να επανέλθουμε σε αυτή τη μεταφορά που αναφέρεται, πρέπει κανείς να αποφασίσει στα 11 ότι θέλει να παντρευτεί το άλλο άτομο όταν γίνει 16. Όταν λοιπόν το έχετε σκεφτεί αυτό το πράγμα, τότε μπορείτε να το προτείνετε στην άλλη πλευρά και να δείτε αν το αποδέχετε. ο κύριο Πώς τώρα. Ευχαριστώ. Ήδη ο Ρούσπεκαν εφέρθηκε σε πολλά από αυτά που ρωτήσατε. Όντω πρέπει να υπάρχει μια επικοδομητική αντιμετώπιση των, των κυρώσεων. Είναι το πιο ισχυρό μέσο που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα έφερε αποτελέσματα. Όμως, συμφωνώ με τον Ρουσμπεκ ότι υπάρχει μεγάλος δυναμισμός μέσα στο Ιράν. Και γιατί και γιατί υπάρχει κακή οικονομική κατάσταση στη χώρα. Οπότε εδώ υπάρχει ελπίδα. Οπότε αυτό που έκανε τα τελευταία χρόνια ο Ρουχανή με τις πιο ριζοσπαστικές ομάδες του πληθυσμού κλπ. ήταν να επανακαθορίσει τα εθνικά συμφέροντα του Ιράν σε σχέση με την διένεξη Ισραήλ-Παλαιστίνης. Ιδίω πρόσφατα όταν είπε ότι οι σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες εξαρτώνται μόνο και αποκλειστικά από τα εθνικά συμφέροντα του Ιράν. Όταν λοιπόν υπάρξει εξομαλισμός με τη Δύση, δεν σημαίνει φιλία, δεν σημαίνει στενές και εντατικέ σχέσεις, αλλά όταν έχει σπάσει το ιδεολογικό ταμπού, μπορούν να γίνουν και τα υπόλοιπα. Και έτσι έρχομαι σε κάτι άλλο που αναφέρατε για τη συμμαχία Σαουδικής Αραβία Ισραήλ. Τα τελευταία τρία χρόνια με το τέλος της αντίστασης μέρος της πολιτικής του Ιράν για το Μεσανατολικό αποτέλεσε στοιχείο επαναξιολόγησης του Ιράν και μας εξέπληξε η αυστηρότητα και η επιτυχία της Αλκάιντα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, πώς έχει επεκταθεί από το Ιράκ στο κέρας της Αφρικής κλπ. Δεν λέω ότι πρέπει να περιορίσουμε το Ιράν τώρα στο στοιχείο των σιτών, παρόλο που έχουν μεγάλη θέση στο σύνταγμα της χώρας. Όμως, χρησιμοποιήθηκε για να επηρεάσει και τις δύο πλευρές. Ήτανε στοιχείο ανταγωνισμού σε δικής ε, Σαουδικής Αραβίας και Ιράν. Και αυτό που θέλω εγώ εδώ να πω είναι ότι με την ίδια λογική το 2001 οι Ηνωμένες είπαν ότι πρέπει να συνεργαστούμε με το Ιράν σε επίπεδο πληροφοριών. Εγώ θα έλεγα ότι στη σημερινή κατάσταση τώρα είναι αναγκαίο αυτό. Παρόλο που παραδέχομαι ότι μόνο μετά αφού έχει κλείσει το πυρηνικό ζήτημα με το Ιράν μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Πάντως είναι σημαντικό να αναλύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πόσο επικίνδυνο είναι το στοιχείο της Αλκαΐντα στην σημερινή κατάσταση. Αλλά γι' αυτό δεν χρειάζεται να μιλήσετε με τους Ιρανούς. Αν πιστεύετε ότι είναι πολύ σημαντικό και γίνεται στρατηγική απειλή πέρα από την τρομοκρατία, πρέπει να συνεργαστούμε με όλου ανεξάρτητα από το τι γίνεται με τα θράπινα δικαιώματα, είτε πρόκειται για το Ιράκ, είτε πρόκειται για το Ιράν, είτε οτιδήποτε. Τώρα για το Ιράκ. Το Ιράν δεν είναι δορυφόρος. Το Ιράκ είναι... έχει τη δικιά του οντότητα. Πλειοψηφία σίτες. Ορισμένοι στην περιοχή όμως αρνούνται την ύπαρξή τους. Είναι ανταγωνιστές μεταξύ τους το Ιράν και το Ιράκ. Γιατί επειδή υπάρχει αυτή η τρέλα της Τεχεράνης, παρόλο που την δεκαετία του 80 όταν ήταν πρόσφυγε στο Ιράν έχει εκπαιδεύσει πολλές προσωπικότητες. Είναι πρώτη φορά που τόσο κοντά δύο δείτε τι γινόταν παλιά, τα προβλήματα που υπήρχαν παλιά στο Ιράν παραμένουν. Υπάρχει πάντα κατάπαυση πυρός, όλα τα ζητήματα της δεκαετίας του 70, του 80, των μειονοτήτων παραμένουν μετά από τόσα χρόνια. Το Ιράν έπαιξε τα χαρτιά του πολύ καλά, δεν μπορεί όμως να επιβάλλει τις απόψεις του στο Ιράκ, πρέπει να διαπραγματευτεί. Τη δουλειά τους την κάνουν πάντως για το συμφέρον τους αρκετά καλά. Τέλος, Ισραήλ σε Δική δεν νομίζω ότι θα υπάρχει συμφωνία, συμμαχία. Υπάρχει κάποια σύγκληση αλλά αν δεν υπάρξει το Παλαιστινιακό κράτος και μια οριστική ειρηνευτική διαδικασία, δεν θα υπάρξει ένταξη του Ισραήλ στην περιοχή, ούτε θα υπάρξουν επίσημα διπλωματικές σχέσεις, για παράδειγμα, ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία. Ιράν και Συρία τώρα, ναι. Το Ιράν δεν έχει εναλλακτική λύση. Plan B. πρέπει να ξέρουμε ότι, πρόκειται, ότι υπάρχει ε, εκεί και στη Βόρεια Συρία και ένα κομμάτι κάπου που ανταγωνίζεται τις ε, Ισλαμιστικές μονάδες και δρούν σαν ένα ανεξάρτητο κράτος, Κουρδιστάν. Και πάλι πάντως πιστεύω ότι από την πλευρά των Ιρανών κρατάνε τα ενία αρκετά καλά στα χέρια τους. Μειονότητες, ναι, για τις εθνικές ε, μειονότητες υπάρχει η πιθανότητα να έχουν φτιάξει αυτήν την υπερταυτότητα του Ιρανού. Διαφορετικά είναι τα πράγματα στο Ιράν για τους Κούρδους από ό,τι είναι στο Ιράκ ή στην Τουρκία. Δεν είναι τόσο εύκολο να επιχειρηματολογήσουμε. Παρόλο που υπάρχουν ιδιαιτερότητες, παρόλο που υπάρχουν αποσχιστές, αυτονομιστές, κινήματα δηλαδή τέτοια, μέχρι τώρα εξακολουθεί η κατάσταση να είναι πολύ μεικτή και δεν βλέπω εδώ να κυριαρχούν οι μεν στους δε. Οι Σουνίτες στο Ιράν είναι ένα από τα επιχειρήματα που ακούστηκαν τελευταία ότι οι συνοστές ε, και άλλοι προσπαθούσαν να, έχουν, ε, να είναι επικεφαλής στην αστυνομία και αλλού. Συμφωνώ. ότι δεν είναι σαφής κατάσταση όσον αφορά τις μενότητες στο Ιράν. Ευχαριστώ, πολύ. Θέλω να σας ε, πληροφορήσω ότι η πρώτη εξέταση των, της σύστασής μας θα γίνει στην Επιτροπή μας στις 10 Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ.